Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I am very glad. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε και πάλι. Μετά την συνάντηση των συντονιστών το πρωί και τις 2,5 ε, ώρες της συνάντησης της Επιτροπής φτάσαμε στην απογευματινή μας συνεδρίαση και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Επίτροπο Κάρλος Μουέδας που πολύ χαιρόμαστε που τον έχουμε μαζί μας για την ανακοίνωση της Κομισιόν για το FP7 ex post αξιολόγηση και σχετική έκθεση. που και για μένα προσωπικά, λέει ο κ. Μπούζεκ, είναι πολύ σημαντική και πολύ χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Η έκθεση για το PP7 υπευλήθη το Νοέμβριο του 2015 και δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο και εμείς ως Επιτροπή Ήτρε είμαστε υπεύθυνοι framework programs starting from the first one until the eighth. Το 8.1 είναι ο Horizon 2020 από τα διάφορα προγράμματα του πλαισίου. Παρακαλώ λοιπόν τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Γέρζη Μπούζεκ, αγαπητά μέλη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι τιμή για μένα που είμαι στην Επιτροπή αυτή για να ανταλλάξουμε απόψεις, για να συζητήσουμε Νομίζω τον Ιούλιο ήταν η τελευταία φορά που ήμουν εδώ και πολύ χαίρομαι που έχω και πάλι την ευκαιρία να σας μιλήσω για την πώς ε, ταξιολόγηση του 7ου πρόγραμμα πλαίσιο FP7 7 χάρην συντομίας. Αυτά ε, ενεκρίθησαν τον Ιανουάριο στις 19, τα διαβίβασα αμέσω στον πρόεδρο Μπούζεκ και σίγουρα θα έχετε λάβει αντίγραφα της ανακοίνωσης για την αξιολόγηση επί του αντικτύπου για την έρευνα και ανάπτυξη που δεν μπορούμε αρκετά να το υπογραμμίσουμε και να το τονίσουμε και για δύο λόγους. Αφενός, η αξιολόγηση αυτή που έγινε με απόλυτη ανεξαρτησία από μια ανεξάρτητη επιτροπή και μας λέει ότι αυτό είναι κρίσιμη σημασία για την οικονομία μας. Το σημαντικό είναι ότι ποσοτικοποιεί δεν είναι απλά ευχές και επιθυμίες, είναι αριθμοί που τους έχει επιβλέψει ο καθηγητής Λουίς Φρέσκο. Είναι θεμελιώδες επίσης για την ευθύνη που έχουμε προς Ευρωπαίους πολίτες, για τη λογοδοσία Η εξελόγηση αυτή λοιπόν θα ληφθεί υπόψη στην επερχόμενη διάμεση εξελόγηση του Horizon 2020 που την περιμένουμε για το 2017 και πιστεύω και ελπίζω να με βοηθήσετε ότι αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ότι θα είναι δηλαδή πολύ σημαντικό, απαραίτητο να έχουμε τις απόψεις σας ή στην προετοιμασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Θα ήθελα αυτό πραγματικά να το κάνουμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα υπογραμμίζοντας κάποια από τα βασικά πορίσματα της αξιολόγησης αυτής, η οποία δείχνει σαφέστατα ότι μέχρι στιγμής το PP7 είχε αντίκτυπο επί των ερευνητών, επί των καινοτόμων, επί της οικονομίας, επί γενικώ της κοινωνίας και δείχνει μια σαφέστατη πανευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το PP7 είχε 55 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικό προϋπολογισμό και αν το σκεφτεί αυτό κανείς προσεκτικά είναι απλώς το 7% των συνολικών δημοσίων δαπανών. Το 70% ήταν για τα πανεπιστήμια το 25 ήταν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και επενδύσεις, εκ των οποίων το ίμιση για τις ΜΜΕ και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Και θα ξεκινήσω από το πρώτο που ήθελα να αναφέρω στα πλαίσια του αντικτύπου του FP7 στους ερευνητές και στην καινοτομία. 170.000 δημοσιεύσεις που οδήγησαν σε γνώση για 1.007 υποβολές ε, αδειών ε, ευρεσιτεχνίας που οδήγησαν σε 7.100 επιχειρήσεις κατόχους αδειών ευρεσιτεχνίας που δείχνει ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δώσει σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτομία. άνω του 70% των αδειών αυτών ήταν open access και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος που να ακολουθήσουμε. Και έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο από τον ευρωαϊκό μέσο όρο. Πιο συχνά δημοσιευόμαστε σε υψηλού κύριους επιστημονικά περιοδικά και μέχρι το 30% των δημοσίευσεων αυτών προκύπτουν από προγράμματα χρηματοδοτούμετα από το PP7 που είναι μεταξύ του 10% των υψηλότερου κύρου επιστημονικών δημοσιευμάτων. Δηλαδή βρισκόμαστε στην αφρόκρεμα, στην υψηλότερη ποσόστοση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί τη βάση αυτών λοιπόν, ο αριθμός των δημοσίευσεων στα επιστημονικά περιοδικά, ο αριθμός των ε, βραβεύσεων Νόμπελ, ε, είχα την ευκαιρία να πάω και στον Ταβός ε, πριν από μία εβδομάδα, μαζί με δύο βραβεία Νόμπελ με χορηγίες του ERC, ο κύριος Νοβόζελοφ και ο καθηγητής Πισαρίδης. Ένας από τους καλύτερους μακροοικονομολόγους στον κόσμο. Μιλούμε λοιπόν για ένα σήμα επιστημονικής αριστείας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να διαβάσουμε στους πολίτες την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την πραγματική θετική επίπτωση στην οικονομία, τις προβολές που έχουμε στη διάθεσή μας, με τις οποίες βεβαίως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά δείχνουν μια τάση, μια πραγματική τάση, ένα θετικό αντίκτυπο. Κάθε ευρώ επένδυσης στο PP7 έχει δημιουργήσει 11 ευρώ μέσω καινοτομιών και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Αυτό μας δείχνει ότι η αυξανόμενη ανάπτυξη είναι περί τα 11 δις το χρόνο. Ε, στα 25 χρόνια 500 δις. Θα δημιουργήσουμε 130.000 νέες θέσεις εργασίας ερευνητών και 160.000 νέες θέσεις έμεσα για τα επόμενα 25 χρόνια. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα νούμερα, αλλά ο αντίκτυπος είναι απολύτως θετικός. Και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το FP7. Και αν δούμε αυτά που κάναμε, είχαμε πέντε κοινέ πρωτοβουλίες ε, τεχνολογίας, ε, καινοτόμα φάρμακα, υδρογόνο, ε, κυψέλες καυσίμου, εταιρικές σχέσεις για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για τα μελλοντικά ενεργειακά αποδοτικά κτίρια του μέλλοντος αλλά σκεφτούμε και το τρίτο που είναι ο αντίκτυπος επί της κοινωνίας, επί των Ευρωπαίων πολιτών σε ένα διάστημα που αντιμετωπίζουμε διάφορες προκλήσεις θεωρούμε ότι το FP7 έχει καταφέρει να θέσει μια κοινή επιστημονική βάση για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις, την στέγαση, την, τα τρόφιμα, την ε, φτώχεια, τον αποκλεισμό, τα περιβαλλοντικά. Περί τα 25,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι ουσιαστικής θεμελιώδους εμεσίας για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της αριστείας στην Ευρώπη. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα εξέταζα εγώ όλα τα, τα έργα αυτά και μερικές φορές δεν λέμε όλη την ιστορία στον κόσμο. Υπάρχει ένα ε, πρόγραμμα που λέγεται SolarJet το οποίο δημιούργησε μια συνταγή για κάψιμο με νερό, διοξείδιο του άνθρακα και ηλιακή θερμότητα. Δηλαδή μετατρέπουμε το διοξείδιο σε πόρο και αναρωτήθηκα, μα πράγματι. Και ανέτρεψα το 2014 που είχαν δημιουργήσει ένα δοχείο κυροζήνης ακριβώς με αυτή την τεχνική. Αυτή, τέτοιου είδους είναι οι αφηγήσει που θα πρέπει να διαβάσουμε στους πολίτες, γιατί αυτές θα αλλάξουν το μέλλον μας. Όσο περισσότερο λοιπόν επιμείνουμε και είμαστε ακριβείς σε αυτές τις περιγραφές, τόσο περισσότερη στήριξη θα έχουμε από τους πολίτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο της επιστήμης και της ε, τεχνολογίας. Άλλος ένα αντίκτυπος του προγράμματος πλαίσιο είναι ο διεθνής αντίκτυπος. Το ονομάζουμε Open to the World. Είχαμε 170 συμμετέχουσες χώρες στο PP7. Ένα πέμπτο των συμμετοχικών προγραμμάτων είχαν συμμετέχοντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδεδεμένες χώρες Α, ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Είχαμε 11 οργανισμούς, 9 περιφέρειες σε 6 χώρε. Υποστηρίξαμε την κινητικότητα άνω των 50.000 ερευνητών σε 140 χώρε. 30% των οποίων ήταν εκτός Ένωση. Σχεδόν το ίμιση των ερευνητών από βιομηχανοποιημένες ευρωπαϊκές χώρες παρέμειναν μετά τη δράση και τη χορηγία στην Ευρώπη. Και αυτό μας βοήθησε να ειδοποιήσουμε τα κενά και τις ελλείψεις που πρέπει να πληρώσουμε. Πέντε συγκεκριμένες συστάσεις εδόθησαν και δεν θα τις διατρέξω όλες καθώς τρέχει και ο χρόνος αλλά μερικές από αυτές ήδη έχουν καλυφθεί μερικώς από τον ορίζοντα 2020. Κάποιες άλλες μας δείχνουν ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα δουλειά. Να σας δώσω τρία από τα παραδείγματα πρωτού ολοκληρώσω. Το FP7 ήταν εξαιρετικά περίπλοκο και δεν επέτυχε ευρεία κλίμακα απλούστευση. Όπω Όπως γνωρίζετε και χάρη στο Κοινοβούλιο, ο ορίζοντας 2020 έχει αναλάβει σημαντικότατα βήματα για τους κανόνες συμμετοχής και τους χρόνους ε, καταβολών ε, και συνεισφορών. Αλλά δεν ήταν επαρκές και πρόσφατα ε, κινήσαμε μια ευρύτατη δημόσια διαβούλευση για να έχουμε εισρωές, input και να προχωρήσουμε με τις απλουστεύσεις. Ήρθαμε σε επαφή με άνω των 5.000 ανθρώπων για να έχουμε τη δική του γνώμη. Χρειάζεται να αυξήσουμε την ελκυστικότητα της Ένωσης για τους ερευνητές και καινοτόμους επιστήμονες και πρέπει συνεχώς να ομαδοποιούμε καλύτερα, να πετυχαίνουμε συνέργειες μεταξύ των πιο καινοτόμων προγραμμάτων. Θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του. Τόσο πολλοί από εσά έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και εδώ στο Κοινοβούλιο διοργανώνουμε, θα διοργανώσουμε πάρα πολύ σύντομα ε, μια συζήτηση ακριβώς για αυτή την καλύτερη οργάνωση όλων αυτών των μέσων και εργαλείων Βεβαίω λέει ο πρόεδρος Μπούζη. Προσπαθούσα λοιπόν να πω ότι πολλοί από αυτούς τους οποίους επισκέφθηκα τις ε, ε, νέες επιχειρήσεις, τις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες μας λένε ότι έχετε τόσα πολλά μέσα αλλά εμείς δεν ξέρουμε πού να πάμε. Η δημιουργία λοιπόν μια ενιαίας θηρίδας είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον μας και μάλιστα ανταποκρίνεται και σε μία από τις συστάσεις της εκθέσεως και επίσης εργαζόμαστε επί της θέσπισης, εφόσον θα είναι καλή ιδέα, αυτού που θα ονομάζουμε European Fund of Funds, δηλαδή νέες γενναίες καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Very, very, very, uh, um, uh, Αυτές λοιπόν είναι οι απαντήσεις, οι απτές και συγκεκριμένες απαντήσεις στις συστάσεις. Επίσης η αξιολόγηση βρήκε ότι οι διαφορετικές πτυχές του PP7 έχουν λειτουργήσει μεμονωμένα και η διαμερισματοποίηση του προγράμματος ήταν υπερβολική. Αυτό βελτιώθηκε μέσω του ορίζοντα 2020 χάρη στην εσφορά σας. Και γι' αυτό αφιερώσαμε όλη την προσοχή μας στο να επιτύχουμε καλύτερες και πιο αποτελεσματικές συνέργειες ε, μεταξύ άλλων και στα διαρθρωτικά ταμεία και έχω πολύ καλά νέα για σας σήμερα γνωρίζετε ότι έχουμε κινήσει ε, αυτό που ονομάζουμε ε, ε, ανώτατο όριο αριστείας μεταξύ των διαρθρωτικών και του ορίζοντα δηλαδή αν υπάρχει ένα έργο, ένα πρόγραμμα επί μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι πολύ καλό αλλά δεν έχουμε επαρκή κονδύλια στον ορίζοντα τότε εμείς θα υπογράφουμε ένα πιστοποιητικό που θα λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτήθηκε αλλά είναι εξαιρετικό. Μέχρι στιγμή, 500 τέτοια πιστοποιητικά έχουμε υπογράψει. Και θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανία και την Ιταλία που υπήρξαν οι ηγέτε, οι καθοδήγητέ σε αυτή την προσπάθεια εξέβριση συνεργειών μεταξύ των δύο πηγών χρηματοδότησης και το οποίο είναι εξαιρετικό. Και αυτό το στοιχείο των συνεργειών με οδηγεί στο τελευταίο για σήμερα, δηλαδή το καθεστώς της υλοποίησης, της εφαρμογή του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις επενδύσει. Η Αμερική Τράπεζα υπολογίζει ότι μέχρι το τέλος του 2015 το FPS οδήγησε σε περί τα 50 δις αναμενόμενες επενδύσεις συνολικά που διαρρούνται σε δύο περιοχές. Ε, υποδομές και καινοτόμα προγράμματα. 42 έχουν εγκριθεί συνολικά και έχουμε και τις συμφωνίες, 84 από αυτές που υπεγράφησαν για 8 περίπου δισεκατομμύρια. Περιμένουμε λοιπόν την παραγωγή εσόδων περί τα 2 δις από την λειτουργία αυτών των προγραμμάτων με βιοπλαστικά, ε, ιατρικές μεθόδους, βιοτεχνολογία, βιοπροϊόντα. Έχουμε, δηλώνουμε ικανοποιημένοι. Ερώτηση. Η απάντηση όχι ακόμα. Είναι ο στόχος μας να επιτύχουμε πολλά περισσότερα. Βεβαίως. Και εγώ σε όλες μου τις εθνείς επαφές προσπαθώ να πείσω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία και έρευνα. Το ΕΦΣΙ μας έχει επιτρέψει να έχουμε 750 εκατομμύρια ευρώ εντός του 2015 που έχουμε χρηματοδοτήσει γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρηματοδοτήσει χωρίς το πλαίσιο αυτό και το ΕΦΣΙ περί τα 420 εκατομμύρια ακόμα θα χρηματοδοτήσει για τα καινοτόμα με ε, εργαλεία του μέλλοντος. Έχουμε πολλές ακόμα συμφωνίες που εκκρεμούν προς ολοκλήρωση και αυτοί, αυτές οι πλεονασματικές επενδύσεις, ε, οι επιπλέον επενδύσεις στην στην έρευνα και την τεχνολογία θα πρέπει να διατευθύνουν στην πραγματική οικονομία. Έχουμε την ιστοσελίδα EIPP, European Investment Portal, που θα δείξει, θα περιγράφει όλα τα έργα τα οποία είναι επενδύσιμα, για να το πούμε έτσι, και θα τα συνδυάζει με τις απαραίτητες δυνατότητες και ευκαιρίες με ιδιώτες και ε, κρατικούς χορηγούς, ώστε αλλά αυτά να καταθίστανται πιο ελκυστικά για τους επενδυτές και να γίνουν πραγματικότητα. Έχουμε και ε, μελέτες, εκθέσεις από πέρυσι, επί των επενδυτικών αυτών προγραμμάτων, με πρόσβαση σε διάφορες επενδυτικές υπηρεσίες, για να αναπτυχθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, του Κοινοβουλίου θα ολοκληρώσω με, ένα κουίπ του Μίλτον Φρίντμαν που είπε ότι ένα από τα μεγάλα λάθη είναι να αξιολογούμε τις πολιτικές τα προγράμματα από τις προθέσεις τους και όχι από τα αποτελέσματά τους. Είπε ο Μίλτον Φρίντμαν. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε καλύτερα στο μέλλον προς το όφελο των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό που αναφερόμαστε ε, στα, στην επταετή περίοδο του 7ου προγράμματος πλαισίου και λίγο παραπάνω θα έλεγα γιατί κάποια project συνεχίζουν να τρέχουν και μετά. Έπρεπε λοιπόν να ενημερωθούμε περισσότερο γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε και την προσέγγιση μας προς ε, την έρευνα και κοινοτομία στο μέλλον. Επομένω, είναι απολύτω ε, απαραίτητο να γίνει ανάλυση του παρελθόντος για να συναγάγουμε συμπεράσματα και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ και να καλασορίσω και το προηγούμενο μέλος της Επιτροπής ε, Ήτρε, την κυρία Ρωμάνα Γιόρνταν, που είναι μαζί μας σήμερα και ήταν μέλος ε, της Επιτροπής Ήτρε για 10 χρόνια. Θεέ μου. Τι θυμόμαστε κάποιοι. Και τώρα η κυρία Ρωμάνα Γιόρνταν είναι επίσημη εκπρόσωπός μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Ήτρε βεβαίως στο Προεδρείο του ΑΙΣΕΡ των Ενεργειακών Ρυθμιστικών Αρχών. Εξαιρετικά σημαντική θέση. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε σήμερα και είστε σε επαφή μαζί μα. Όπως και άλλα πρώην μέλη της Επιτροπής μας. Ας ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Έρλερ, εισηγητής αλλά και εκπρόσωπο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και εισηγητής για τον ορίζοντα 2020. Στα αγγλικά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχικό, αρχικός να σας πω ότι και ο Τζέρζι Μπούζεκ ήταν εισηγητής για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, επομένω ε, τα γνωρίζει πολύ καλά και γνωρίζει και αυτές τις επιτυχίες που αναφέρατε. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή, ε, μπορούμε να μιλούμε και για τις επιτυχίες, αλλά η ανάλυση των όσων ε, βλέπουμε εδώ μπορεί να μας δώσει και μια ιδέα για το μέλλον. και μπορούμε να εξετάσουμε και ζητήματα που προκύπτουν από την ε, αναθεώρηση και την επανεξέταση του 7ου προγράμματο πλαίσιο. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπόθηκαν πολλά για συνέργειε ε, και τη μόχλευση. Ίσως είναι στο χαρακτήρα αυτό του 7ου προγράμματο πλαίσιο. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και, η ανάλυση του εισηγητή έδειξε ότι υπήρχαν ελλείψεις σε τη φορά της συνέργειες με άλλα κονδύλια και ταμεία, αλλά και σε ό,τι φορά την μόχλευση που είχε άμεση σχέση με τον 2020 και με το ΕΦΣΥ, αλλά βλέπουμε ότι κάπως αποφεύγουμε αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του FP7. Μετά το δεύτερο το οποίο ήθελα να θίξω είναι το χάσμα καινοτομίας. Μία από τις ελλείψεις και αδυναμίες του FP7 είναι και πάλι ο κατακαιρματισμός μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 13. Πρέπει για την ενδιάμεση αναθεώρηση να το εξετάσουμε περισσότερο αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στον του 2020, όμως παραμένει αυτό το ζήτημα πολύ σημαντικό και πάντα υπήρχε συνένεση μεταξύ των 15 και των 13 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι δεν βλέπουμε αν στον άλλον έτσι, ότι εξακολουθεί να κυριαρχεί η έννοια της αριστείας στο πρόγραμμα. Και αυτό μας υποχρεώνει ακόμη περισσότερο να εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να επανισορροπήσουμε περισσότερο μέσω της ενδιάμεσης αναθεώρησης το πρόγραμμα αυτό. Και κάτι τελευταίο, που είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου για την ανάμεσα αναθεώρηση είναι η μέτρηση. Μία από τις αδυναμίες της ανάλυσης του FP7 οφείλεται στο γεγονός ακριβώς που, στον τρόπο μάλλον που έχει σχεδιαστεί. Είναι στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε και μετράμε ε, τις, τα διπλώματα και τις δημοσιεύσεις. Όμως ο Horizon 2020 ακριβώς έχει σκοπό ε, να αντιμετωπίσουμε ακριβώς ε, τις προκλήσεις που έχουμε ενεργειακή απόδοση ή εκπομπέ του του άνθρακα. Και αυτό όμω οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο μέλλον δεν θα πρέπει να μιλούμε μόνο για τους αριθμούς, ε, για τα διπλώματα τεχνία και το καθεξή, αλλά σε έναν βαθμό να εξετάζουμε και τι ακριβώς συνιστά επιτυχία. Αν δείτε για παράδειγμα την πρόκληση των τομέα τη ενέργεια, το ζήτημα δεν είναι μόνο ο αντίκτυπο επί συγκεκριμένων στοιχείων, αλλά και το κατά πόσο έχουμε πετύχει έναν στόχο. Για τη μέτρηση λοιπόν θα μπορούσαμε να λέμε ότι έχουμε προσδιορίσει έναν στόχο από τεχνολογική σκοπιά για την μείωση των εκπομπών του άνθρακα, το αναφέρω επί παραδείγματι, αλλά μετά πρέπει να πούμε ορίστε τα αποτελέσματα, ενδεχομένω να προβλέπονται και άλλα ε, στοιχεία για συνεχιζόμενα προγράμματα, αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν διαφοροποίηση, γιατί και από τη φύση του ο ορίζον 2020 διαφέρει από το FP7 και γι' αυτό θέλω να δω κατά πόσο αυτό έχει ληφθεί υπόψη στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Βεβαίω περιπλέκει και την ίδια την αναθεώρηση, όμως είναι απαραίτητο στοιχείο για να κατανοήσουμε πόσο επιτυχής μπορεί να είναι αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ, Χριστιαν, λέει Εκ μέρους των σοσιαλιστών, συνάδελφε Σωρίνιο. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ελπίζω να μην ε, έχει πρόβλημα να μιλήσω τη μητρική σας και μου γλώσσα. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα εδώ σήμερα και σα ευχαριστώ και για την ε, παρουσίαση της αξιολόγηση του 7ου Προγράμματο πλαίσιο που δείχνει και πάλι πόσο σημαντικό είναι να εξετάζουμε την ε, πολιτική σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Μπορούμε ε, να αξιολογήσουμε και αυτή την ανάλυση. Το σημαντικό είναι να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή τη διαδικασία τι μας προσφέρει αυτό. Ξέρουμε ότι η έρευνα, η γενοτομία, η επιστήμη είναι κρίσιμη σημασία στοιχεία για την καταπολέμηση των προβλημάτων προκλήσεων που έχουμε στον πλανήτη μας. Και όλα αυτά η έρευνα και η ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες ε, μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και άλλες προκλήσεις όπως είναι η εκπομπή του διευθυντήτου του άνθρακα. Χρειάζεται λοιπόν και νομική αντιμετώπιση, αλλά και τεχνολογική και επιστημονική. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε και τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις ε, για να προβάγουμε τους ε, στόχους μας. Και σε αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές θα μπορούσε κανείς να αναφέρει, αλλά αφορούν κυρίως και συνδέονται και με τα κονδύλια που διατίθενται για την επιστήμη και την ανανέωση. Αναφερθήκατε κύριε Επίτροπε για ε, την έγκριση των προπολογισμών για το πρόγραμμα Juncker. 50 εκατομμύρια αναφέρατε από το ΕΦΣΙ, χρήματα που έχουν ήδη ε, διαδοθεί, διατεθεί, όμως μιλούμε για μεγάλα έργα. Μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικά έργα, χωρίς όμως να είναι μεγάλα σε κλίμακα για τον ορίζοντα 2020, τότε το, σε αυτή την περίπτωση του προγράμματος ορίζον 2020, το ε, σχέδιο Juncker είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν υπάρχει ακόμα εκεί η θηρίδα. Είναι κάτι απαραίτητο όμως. Χρειαζόμαστε άμεση πρόσβαση. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά μικρής κλίμακας έργο. Πρέπει να διασφαλιστεί και αυτό. Δεύτερον, η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα. Στην Ευρώπη υπάρχει κατακαιρματισμός ε, και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα δεν μας επιτρέπουν άμεση πρόσβαση, για παράδειγμα, και σε επιστημονικά δεδομένα. Πολλές φορές ξέρουμε ότι υπάρχει ε, διπλή χρηματοδότηση, αλλά πολύ κακή πρόσβαση σε δεδομένα. Τι θα κάνετε για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και τέλος, κάτι ακόμα, σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό ε, και την αντιμετώπιση ε, του ψηφιακού χάσματος μεταξύ ε, Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Είναι πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε, γιατί και εγώ είμαι αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας με τη Βραζιλία. Πήγα και στη Βραζιλία, στο Μελεζόντα και εκεί είδα ότι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού υπάρχουν μεγάλε υποδομέ. Είναι λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να είστε σε θέση να μας πείτε μερικά πράγματα παραπάνω για τα πρακτικά αυτά παραδείγματα. Ευχαριστώ κύριο Στοσενόφσκι. Έχει το λόγο εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών. Θα μιλήσω κι εγώ τσεχικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα όσα μας ανέφερε σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Με ικανοποίηση βλέπουμε όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία γιατί είναι σημαντικό για μας όταν έχουμε την εκκίνηση του ορίζοντα 2020 να έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι είναι σημαντικό με ανεξάρτητο τρόπο να καταρτίζονται αυτά τα προγράμματα. Ίσως παρέλειψα μία πληροφορία. Θυμάμαι ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο συμπεριλάμβανε επίσης προσδοκίες και σε ό,τι αφορά την εξολόγηση αντικτύπου. Πώς όμως ανταποκρίνονται αυτές ε, οι προβλέψεις με τα πραγματικά, πραγματικά αποτελέσματα της αξιολόγησης. Αυτό θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε προβλέψεις ε, και στο μέλλον. Και θα ήθελα να σχολιάσω τα είπα συνάδελφος προηγουμένως ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο πολλές φορές ε, σχολιάστηκε εδώ στην Επιτροπή μας με πολύ διαφορετική χρηματοδότηση στις επιμέρους ε, χώρες. Αν είσαι για τρει-τέσσερι χώρε, θα μπορούσε να είναι τοπικό το ζήτημα. Αλλά 13 στου 28, αυτό φαίνεται να δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά είτε στις συγκεκριμένες χώρες, χώρε, κράτη-μέλη, είτε δεν ακολούθησαν το σύστημα όπως πρέπει, Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε. Γνωρίζουμε ότι το σύστημα του 7ου πρόγραμμα πλαίσιο, πλαίσιο ήταν πολύ σύνθετο ό,τι αφορά την παρουσίαση και υποβολή των έργων. Για εμάς αυτά τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά, ιδίω στον επιστημονικό τομέα, σε σχέση και με τα διαφορετικά ταμεία, ούτω ώστε να μην αποκλείονται συγκεκριμένα κράτη-μέλη Ευχαριστώ και πάλι. Αναφερθήκατε στο 85% ε, που δόθηκε στα παλαιότερα των κρατη κράτη-μέλη και το υπόλοιπο στις λεγόμενες νέες χώρες, αλλά βέβαια τόσο νέες δεν είναι πια. Είναι όμως χαρακτηριστικό. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, εκ μέρους της ΓΚΟΕ, η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα που ήρθατε εδώ να συζητήσουμε ακριβώς ε, την εξπόστ αξιολόγηση του προγράμματος πλαίσιο. Έχω ορισμένες παρατηρήσεις γιατί κάποια στοιχεία νομίζω ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν την αξιολόγηση. Αναμφίβολα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα επενδύσεων. Όμως, εξετάζοντα μάλλον την ε, αξιολόγηση, την έκθεση αξιολόγηση, περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια όλοι οι ενδείξεις και ότι συμμετέχουν με ασύμετρο και άνισο τρόπο τα 27 και 28 κράτη-μέλη, αλλά συνολικά αφορούσε πολύ περισσότερες χώρες, 117. Από εκεί πέρα βλέπουμε και την συμβολή αυτού του προγράμματος ε, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Δεν είναι τέλεια βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, είναι σημαντική και η τεχνολογία για την ανάπτυξη ε, σε κάθε κοινωνία. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έχει επιληθεί ούτε από το 7ο πρόγραμμα πλάσιο ούτε από τον ορίζοντα 2020. Όλα ένα και συχνότερα ε, μιλούμε για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά για το τι είδου απασχόληση αυτό δεν το εξετάζουμε. Βλέπω λοιπόν στην έκθεση εξολόγησή σα ότι και κρίνω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό, τότε θα έχουμε και πάλι και στον ορίζοντα 2020 αυτό το ζήτημα. Ανάπτυξη τώρα, απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά το θέμα είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος που εργάζεται σε αυτά τα προγράμματα ε, εργάζεται από καθεστώ επισφάλεια. Δεν έχει μια αξιοπρεπή θέση εργασία και δεν είναι αυτό το μοντέλο το οποίο εμεί επιθυμούμε για την ε, δημιουργία θέσεων εργασία. Επομένω, δεν επιλύεται αυτό το ζήτημα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και βλέπουμε ότι και τώρα που βρισκόμαστε στην αρχή του 2020, το ίδιο διαπιστώνουμε. Επομένω, κύριε Επίτροπε, πώ μπορούμε να εξακολουθήσουμε να εξετάζουμε το ζήτημα τη ε, ανάπτυξη και τη απασχόληση όταν η πλειονότητα αυτών των εργαζομένων τελούν υποκαθεστώς ε, επισφάλειας και απόλυτης αβεβαιότητας. Και μάλιστα μιλούμε για άτομα με πολλά προσόντα, ιδιαίτερα καταρτισμένους. και, δεν, και μάλιστα εξαρτάται το μέλλον αυτού του προγράμματος από όλα αυτά τα άτομα που δεν έχουν λάβει καμία εγγύηση για το μέλλον τους. Και όταν μιλούμε για ανάπτυξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξουν μεγάλες ε, επενδύσεις. Δεν είναι ένας από τους ε, βασικότερους πυλώνες, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη εκτός και αν καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για αυτό το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, να τους διασφαλίσουμε τα βασικά δικαιώματα σε μια ασφαλή και σίγουρη θέση εργασίας. Επομένω, για το FP8 και το 2020, σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε, ούτω ώστε αυτοί οι άνθρωποι να δίνουν τον καλύτερο του σε αυτό και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πούμε κάποια στιγμή ότι έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπολείπους. Ευχαριστώ πολύ ε, για τις παρατηρήσεις σας. Η κυρία Κάπελ, ε, εκ μέρους του ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο για την παρουσίασή του. Σας αρέσει να έρχεστε στο κοινοβούλιο και σα βλέπω αρκετά συχνά σε συνεδριάσεις. Ε, και είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το ότι δείχνετε τόσο ενθουσιασμό για την έρευνα και καινοτομία. Είναι τομεί εξαιρετικά σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη τη, γιατί είναι μοχλό ε, ανάπτυξη και απασχόληση. Και πρόκειται για μέτρα, για προγράμματα τα οποία χρειαζόμαστε επιγόντω για να υπάρξει ανάπτυξη. Τώρα, Μιλήσατε για τον βασικό αντίκτυπο του 7 προγράμματος πλαίσιο και πρέπει να αναφέρω ότι τα επιτεύγματα είναι εντυπωσιακά. Και μάλιστα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα του κόσμου με 55 δισεκατομμύρια ευρώ. 25 ερευνητικά προγράμματα σημαντικά και δεν έχουν ολοκληρωθεί καν και εξακολουθούν και εργάζονται οι ερευνητές σε αυτά. Η έμεσες επιπτώσεις, στη μόχλευση δηλαδή του 1 ευρώ στα 11 ευρώ και οι 92.000 πρόσθετες εργασίες οι οποίες θα ξεπηδήσουν από αυτά τα προγράμματα για τα επόμενα χρόνια καθώς και μια δημιουργία αξία τη τάξη των 500 και δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά είναι τρομερά εντυπωσιακά και δείχνουν πόσο σημαντική είναι η έρευνα και η ανάπτυξη για την οικονομία και για του ανθρώπου εν τέλει στην Ευρώπη. Όπως είπατε κι εσείς, το πρόγραμμα πλαίσιο 7 ήταν διεθνές, με συμμετοχή ερευνητών από 170 χώρες. Και μόνο στο πρόγραμμα Marie Curie ήταν 50.000 ερευνητές από πολλές δεκάδες χώρες. Αυτό που μου άρεσε επίσης ήταν, και το είπατε σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις, ότι έχετε δημιουργήσει task force για την πολιτική στήριξη. Έρευνα και ανάπτυξη είναι από τους μεγάλους στόχους μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 3% του ΑΕΠ να αποδίδει η έρευνα και ανάπτυξη. Και από τις πρόσφατες φθινοπορεινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες μέλη δεν είναι τόσο επιτυχημένες, δεν φτάνουν δηλαδή ούτε μακράν το 3%. Βρίσκω λοιπόν λογικό αλλά και ρεαλιστικό να πάτε επί τόπου και να χορηγήσετε συμβουλές για το πώς μπορούν να ξεκινήσουν μια προσπάθεια ώστε να, είναι, να αποδειχθούν πιο επιτυχημένοι για να επιτύχουν το 30% του 2020. Ελπίζω ότι και στο το 2020 θα μπορέσει να ληφθεί αυτό υπόψη, δηλαδή ένας βελτιωμένος συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων. Βελτιωμένος συντονισμός με τις ευρωπαϊκές συστάσεις, δομές, επενδυτικές δομές. Ήταν λοιπόν το πρόγραμμα πλαίσιο 7 που λιγότερο ήταν ωστόσο στοχευμένο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τη startup. Θα δούμε και στο τέλος του έτους τι θα αποδώσει το νέο πρόγραμμα μιλούν για μια μόχλευση της τάξης του 1 προς 12. Κάτι που πρέπει να σημειώσει κανείς ακόμη είναι η διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στο παγκόσμιο επίπεδο. Τα 80 δισεκατομμύρια για το νορίζοντα 2020 είναι πολλά. Αν δείτε όμως τι κάνουν χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα ή και οι Ηνωμένε Πολιτείες θα δείτε ότι οι δημόσιες ταπάνες τους για την έρευνα και ανάπτυξη είναι πολύ ψηλότερες από αυτές της Ευρώπης. Και πιστεύω, αλλά το είπατε κι εσείς, ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε ο τομέας αυτός που είναι πραγματικό θερμοκήπιο για την ανάπτυξη να συνεχίσει να στηρίζεται και να προωθείται. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ε, όπως βλέπετε λοιπόν ή όπως ακούσατε ο πρώτος γύρος ερωτήσεων κύριε Επίτροπε των πολιτικών ομάδων και τώρα σας παρακαλώ να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα απαντήσω πρώτα πορτογαλικά, αν δεν έχετε αντίρρηση, για να απαντήσω στον Ευρωβουλευτή, τον οποίο επιθυμώ να συγχαρώ κιόλα στην Ευρωβουλευτή, μάλλον την κυρία Μαρίζα Ματίας και στον άλλο συναδελφό μου βεβαίω από την Πορτογαλία. Κυρία Ματίας συγχαρητήρια πρώτα πρώτα και για τα αποτελέσματα της προεδρικής εκλογής στην Πορτογαλία. Ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη η εκστρατεία σας και ιδιαίτερα θετική η θέση σας, η τοποθέτησή σας. Πραγματικά, στο το καπέλο. Τώρα για το θέμα. Αυτό που φίξατε είναι γενικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Και τέτοιο το οποίο βλέπουμε στην αγορά εργασίας και που ξεφεύγει από τα καθαρά πλαίσια της οικονομίας, της ε, καινοτομίας, ένας, ε, ε, ένα ολόκληρο τμήμα του πληθυσμού, όλο και νεότερο. Έχει θέσεις απασχόλησης που δεν είναι ασφαλείς, είναι λιγότερο προστατευμένες από άλλα τμήματα του πληθυσμού. Εδώ βεβαίω πρέπει να βρούμε λύσεις. Καλούμεθα να βρούμε λύσεις και αυτές οι λύσεις σημαίνουν την ουσία ότι θα επιτύχουμε και μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Έχουμε τις συνθήκες πλαίσια, δηλαδή ορίζον 2020, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Αυτά έχουν το στόχο να γίνει η Ευρώπη πλέον καινοτόμος, πλέον παραγωγική, πλέον ανταγωνιστική και επομένως να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να φροντίσουμε ώστε η νέα γενιά του εργατικού δυναμικού να μπορέσει να απασχοληθεί με καλύτερες συνθήκες. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο οι θέσεις απασχόλησης. Φτιάξαμε και υποτροφίες για τους ερευνητές. Αλλά ε, δεν είναι το μόνο που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και στα πλαίσια της πρόθεσης της καινοτομίας. Εξετάσαμε κατά πόσο η προσπάθειά μας οδήγησε σε δημιουργία απασχόληση τη επιχειρήση εκείνε οι οποίε έλαβαν στήριξη σε σύγκριση με εκείνε που δεν έλαβαν. Αυτέ που έλαβαν χρηματοδότηση όντω όντως, δημιουργήσαν θέσει εργασία. Είναι ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και πάντω τέτοιου αναλύσει θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Για να δούμε και αν αυτέ οι θέσει απασχόληση είναι βιώσιμε. Και αυτό θα είναι μια από τις πιο σημαντικές μας ενασχολήσεις και για να μπορέσουμε να δούμε εάν πραγματικά μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες απασχολήσεως και αν μπορούμε στο μέλλον να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη Ευρώπη της απασχόλησης. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο βέβαια είναι προχωρημένο πλέον. Ο ορίζον 2020 προσεγγίζει. Άλλες χώρες έχουν προχωρήσει περισσότερο, άλλες λιγότερο. Τα κέντρα διάδοση της τεχνολογίας έχουν αποδώσει. Έχουμε και τις διαδικτυώσεις εταιρικών σχέσεων και στην Πορτογαλία. Στην Πολωνία επίσης σημειώσαμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες. επιτυχίες. Η συντηγή του μέλλοντος πρέπει ωστόσο να αναζητηθεί στις συνέργειες μεταξύ ορίζοντα 2020 και διαφορετικών ταμείων. και αυτά τα Centers of Excellence πρέπει να στηριχθούν ακόμη. Θα συνεχίσω βέβαια στην πορτογαλική γλώσσα γιατί έλαβα ερωτήσεις και από έναν άλλο ε, Πορτογάλο Ευρωβουλευτή. Κύριο Ζουρίνιο, αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε πάντα μια ενεργό στάση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτά να εξελιχθούν υποθετικό πρόσημα και τα διάφορα έργα να εκτελούνται επιστημονικά σωστά. Γνωρίζετε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων μου περιλαμβάνεται και η ανοιχτή επιστήμη. Ανοιχτή επιστήμη, έτσι το λέμε εμείς. Ανοιχτή επιστήμη για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν εδώ τρία σημαντικά θέματα. Αφενός, ανοιχτός χαρακτήρα των δεδομένων δημοσιοποίησή τους. Δεύτερον, η ακαιρότητα της ε, επιστήμης. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα, τον ε, ανοιχτό χαρακτήρα των δεδομένων, εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Δύο των οποίων επίκειται η λύση, πρόκειται αφενός για την υποδομή και δεύτερο το copyright. Άρα και τρίτο, υπάρχει και το ζήτημα του επιχειρηματικού μοντέλου. Πρώτα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το υπόδειγμα, δηλαδή πληρωμή για να μπορεί κανείς να αναγνώσει ένα κείμενο. Αυτό είναι μια μεγάλη ε, προσπάθεια που κάνουμε μαζί με την Ολλανδική Προεδρία. Χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα εδώ στην Ευρώπη. Υπάρχει μάλιστα και μια αναφορά ώστε, που ζητεί και μάλιστα έχουν συγκεντρωθεί και άνω των 10.000 υπογραφών από επιστημονικούς κύκλους για να υλοποιηθεί αυτή η δωρεάν πρόσβαση σε έγγραφα. Το οριζόντας 2020 θα, θέλουμε, θα θέλαμε να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ότι θα υπάρξει επικαιροποίηση, update δηλαδή, του δικαιώματος της διανοτικής ιδιοκτησίας, του copyright. Και ε, θέλουμε να προβλέψουμε εξαίρεση σε αυτό το text και data mining, την εξόριξη των εισαγωγικών δεδομένων από κείμενα, εφόσον εξυπηρετούνται επιστημονικοί σκοποί. Οι Ευρωπαίοι επιστήμονες χρειάζονται υποδομές Εγώ συνεργάζομαι με τον συνάδελφό μου για να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό science cloud, νέφος της επιστήμης, όπου εκεί θα μπορούν να προσφεύγουν οι επιστήμονες και να αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αμεσότερη η πρόσβαση. Και η καλωδιακή διασύνδεση με την Λατινική Αμερική είναι τμήμα αυτή τη προσπάθεια. Από την δική μα πλευρά δηλαδή, από την πλευρά τη Κομισιόν, ο δρόμο είναι ανοιχτό. Βέβαια, πρέπει να μπει στη μέση και ο ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί να τα αναλάβει μόνο, στο δημόσιο τομέα όλα αυτά. Όταν θα έχω πληροφορίε για την πρόοδο του έργου, θα σα τι ε, διαβιβάσω αμέσω. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Είναι αυτό ο αυτοκινητόδρομο των δεδομένων, όπω είπατε κι εσεί. Τονίσατε δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η σημασία του έργου και πώς το βλέπουν και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ε, τώρα κύριε Πρόεδρε θα επιστρέψω στην Αγγλική για να απαντήσω στους άλλους συναδέλφους. Έβαλα τους δύο Πορτογάλους σε πακέτο, μιας και ήταν δυο η κυρία Ματίας και ο κύριος Ζωρίνιο. Και μου φάνηκε θα ήταν πιο εύκολο έτσι. Τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Και για την πρώτη ερώτηση, κύριε Έλερα διεπίστωσα ότι δεν κάθεται στη σωστή του θέση γιατί έχει άλλο καρτελάκι μπροστά του. Έτσι δεν είναι. Α, ακριβώ μπροστά του είναι, ναι, το σωστά μας. Ε, για τα σχόλια του κ. Έλερ, συμφωνώ με τα σχόλια αυτά για την μέτρηση του ε, κενού καινοτομίας και το καθεξής για τις μετρήσεις αυτές συμφωνώ μαζί σας Έλερ ότι μετρούμε μονάχα τις ευρεσιτεχνίες και τις δημοσίευσεις. Αυτό με απασχολεί πολύ διότι στον κόσμο που έχουμε σήμερα με τέτοιο πλήθος δεδομένων χρησιμοποιείται αυτά τα δύο benchmark μόνο τότε πάει να πει ότι δεν κάνετε σωστή δουλειά και πάει να πει ότι δεν δίνεται τα σωστά κίνητρα. Μιλήσαμε και για το γεγονό ότι στην Νότιο Κορέα πάνω από 100 επιστήμονες προσκλήθηκαν διότι είχαν αντιγράψει. Καταγγέλθηκαν αυτοί η ειχαν Είχαν αντιγράψει, είχαν κάνει copy-paste. Αυτά είναι βεβαίως πολύ αρνητικά για την ε, επιστημονική κοινότητα. Εγώ πιστεύω με, ότι με όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα και σε ό,τι αφορά την έρευνα και σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα 2020 ότι μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία αυτή και μπορούμε να προσφέρουμε διαφορετικά κίνητρα και στους επόμενους μήνες θα αναπτύξω το θέμα αυτό περισσότερο. Μόλις έλεγα στην κυρία Ματίας ότι μια από τις ιδέες που μας απασχολεί σε σχέση με το έργο Ευρωστάρ είναι να βρούμε την διασύνδεση μεταξύ των επενδύσεων, των χρηματοδοτήσεων και τη δημιουργία απασχολήσεω. Τώρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά είχαμε κάνει τότε για το ευρωστά. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από το να εξετάζουμε μονάχα τι πατέντε και τι δημοσίευσει. Και αν δούμε τι πατέντε σήμερα, θα δούμε ότι είναι μέρο μόνο τη διανοητική ιδιοκτησία. Έχουμε λοιπόν και άλλου τρόπου για να μετρήσουμε τα πράγματα αυτά και νομίζω ότι αυτό θα πράξω και στο προσεχέ μέλλον, δηλαδή θα προτείνω διαφορετικές λύσει και ευχαρίστω θα ακούσω και τι απόψεις σας, τις προτάσεις σας. Όταν μιλείτε τώρα για EU15 και EU13, θέλουμε και να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά ένα από τα πράγματα που έχω αντλήσει από την έκθεση είναι ότι δείχνει ότι υπάρχει αισιοδοξία, διότι και στο PP7. Βλέπετε 13 χώρε μέλη, αυτές που πήγαν δηλαδή από το 2004 και μετά, έλαβαν κατά μέσο όρο 30% περισσότερα ανά εκατομμύρια ευρώ που ε, δαπανήθηκαν σε έρευνα και ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο ακόμα και πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, η σφραγίδα υπεροχή, seal of excellence και αυτές οι συνέργειες με αυτές τις ιδέες μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα σε, α, για τις χώρες αυτές που βρίσκονται ακόμα χαμηλότερα στην κλίμακα. Αυτό το σύλλογο of ήταν μια καλή ιδέα. Είδα προ λίγων ημερών ότι έχουμε υπογράψει πάνω από 500 πιστοποιητικά. Αυτό είναι διότι υπάρχει έλξη για την ιδέα αυτή. Υπάρχει μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον για την ιδέα αυτή. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει περισσότερη προσπάθεια. Και μιλήσατε και για τις συνέργειες τις οποίες είχα αναφερθεί και εγώ και για το κενό καινοτομία που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι στην ενδιάμεση επανεξέταση όπως είπατε και εσείς θα πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο αυτό το θέμα και ελπίζω <clears throat> εκεί να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πλέον καινοτόμες λύσεις για τον κύριο Τασενόφσκι σας ευχαριστώ βεβαίως για τις απόψεις που εκφράσατε σχετικά με τις προσδοκίες για το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Η έκθεση είναι σαφής ότι κάπως οι περισσότερες προσδοκίες ξεπεράστηκαν. Υπερεύημεν τις προσδοκίες δηλαδή σε πολλά σημεία. Και έτσι αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι η απόδειξη ότι όντω δημιουργήθηκαν απασχολήσει, ότι όντω δημιουργήθηκαν, ιδρύθηκαν καινοτόμε επιχειρήσει, ότι, ότι όντω βελτιώθηκε η έρευνα, διότι δόθηκαν τα χρήματα βασισμένα σε αυτήν την excellence. Και το Σενάφσκι επίση μιλήσατε για τα διαρθωτικά ταμεία και τι συνέργειε μεταξύ των. Όπω είπα και στον κύριο Έλερ, χρειαζόμαστε όντω περισσότερε καινοτόμε ιδέε για τη δημιουργία τέτοιων συνεργειών για μεγάλο διάστημα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε συνέργειες εκ των κάτω. Τώρα προσπαθήσαμε να φανούμε καινοτόμοι και να το κάνουμε εκ των άνω, βάζοντας την Επιτροπή να υπογράφει πιστοποιητικά, ελπίζοντας ότι αυτό θα δώσει μια νέα δυναμική στη συνεργασία των ταμείων. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε όντως να προωθήσουμε καλύτερες ιδέες και ελπίζω να με βοηθήσετε σε αυτό. Ερώτηση της κυρίας Κάπελ αλλά δυστυχώς δεν την βλέπω πλέον. Την ευχαριστώ πάντως, ας εγγραφεί στα πρακτικά για τα σχόλιά της. Αναφέρθηκε επίσης στις συνέργειες και στην ανταγωνιστικότητα. Τώρα για την ανταγωνιστικότητα. Ένα από τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης του FP7 είναι ότι έχουμε ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματά του στην οικονομία και οι αλλαγές που βλέπω στα μακροοικονομικά που ασχολούνται με την παραγωγικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου αλλά δεν ασχολούνται ποτέ με την παραγωγικότητα την πολύ παραγωγική παραγωγικότητα είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί αυτό γι' αυτό στα μακροοικονομικά εξετάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου γιατί είναι πράγματα πιο εύκολα να μετρηθούν. Αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι οι χώρες που τα πάνε καλύτερα είναι αυτές που έχουν και περισσότερες πολυσχηδείς, περισσότερο πολυσχηδή παραγωγικότητα. Αυτή δηλαδή που βασίζεται και στην καινοτομία. Και αυτή είναι που δημιουργεί εν τέλει αύξηση και απασχόληση. Αυτή η πολυπαραγωγική παραγωγικότητα είναι αυτή που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε καλύτερες και περισσότερες δουλειές και να σας ανεβάσει στο ανταγωνιστικότερο επίπεδο. Σαν να μου φαίνεται ότι απάντησα σε όλους. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω απαντήσατε σε όλους και όλες. Τώρα να έρθουμε στους επόμενους ομιλητές. Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έβδομο πρόγραμμα απέδωσε πολλά αποτελέσματα. 170.000 δημοσίευσεις μεταξύ άλλων. Ε, Επιπέδου παγκοσμίου ποιοτικά. Αυτές τις 170.000 δημοσίευσεις πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε καλύτερα για την παραπέρα εκπαίδευσή μας. Στην ΣΤΟΑ έχουμε αναπτύξει μια νέα στρατηγική silo and pipes strategy, έτσι λέμε. Πρόκειται δηλαδή ε, φανταστικά για σωλήνες που συνδέουν τα διάφορα σιλό. Μπορεί κανείς να μετρήσει καλύτερα με τα κοινωνικά δικτύα ποιες είναι οι ισροές και οι εκροές από τα, από τα διάφορα, από τους διάφορους τομείς. Ο τομέας ε, Science Matrix λειτουργεί όλο και καλύτερα. Ε, καταβάλουμε προσπάθειες τώρα ώστε αυτά να μεταφερθούν και στην παιδεία ξεκινώντας από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, αλλά και στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις ή και στους μεγάλους ομίλους. Νομίζω ότι είναι σωστό επίσης, και εσεί το είπατε, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στόχευση στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. 17 project από την ενέργεια Χρηματοδοτήθηκε μάλιστα ένα έργο με 714 εκατομμύρια. Εάν το συγκρίνω με το πρόγραμμα Eurostar, έλαβε πολύ λιγότερα και τα 17 από τα 17 project στην ενέργεια μόνο λίγα ήταν μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ χρειάζεται λοιπόν να καταβληθεί εντονότερη προσπάθεια. Έχουμε και το project τώρα Performance Based Budgeting, εγγραφή στον προπολογισμό στην βάση της απόδοσης και αυτά θα τα μετρήσουμε και στην βάση της απόδοσης σε απασχόληση, σε παραγωγή ΑΕΠ, αλλά και σε φορολογία, διότι θέλουμε να ταΐσουμε καλά την αγελάδα την οποία μετά θα αρμέξουμε. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε να έχουμε υπόψη μας ως μέτρα. Ευχαριστώ. Κουντρίτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπη, αναφέρθηκε εδώ ότι έχουμε μια, ένα κενό μεταξύ των 15 και των 28 κρατών μελών ως προς τη χρηματοδότηση εντός του PP7 και πρόκειται για μια δραματική διαφορά, ένα τεράστιο κενό. Και εντός του σχεδιασμού του ορίζοντα 2020 είχε συμπεριληφθεί ένας μηχανισμός ώστε να βοηθηθούν τα νέα κράτη-μέλη, τα μετά το 2004, να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο αριστείας. Και εσείς είπατε, μιλήσατε για ένα συνδυασμό χρηματοδότησης από τον ορίζοντα και από τα θεωρητικά. Και ότι αυτή θα ήταν η συνταγή ενίσχυσης της αριστείας στα νέα κράτη-μέλη. Όμως, αναφέρθ, αναφερθήκατε στο σήμα αριστείας αλλά η χορήγηση του σήματος αυτού εξασφαλίζει ότι το αντίστοιχο έργο στο οποίο θα χορηγηθεί το σήμα αυτό θα εξασφαλίσει η χρηματοδότηση. Επίσης αυτά τα προγράμματα twinning και teaming που επίσης προέρχονταν για τη χρηματοδότησή τους από τα διαρθρωτικά και τον οριζόντα. Και εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, αυτή είναι η μόνη δυνατότητα και ευκαιρία για τα ταμεία που έχουν οριστεί, προβλεφθεί για επιστημονικής αριστείας έργα να μην χρησιμοποιηθούν για χαμηλότερης ποιότητας έργα και προγράμματα. Επομένως, η ερώτησή μου είναι, έχετε κάποια άλλη νέα πρόταση, εκτός από αυτό το σήμα χρηματοδότησης, ε, αριστείας με συγχωρείτε, για τα teaming και twinning, γιατί είναι η μόνη ευκαιρία όπως μου φαίνεται, ε, να βελτιώσουμε την κατάσταση και να βελτιώσουμε συνολικά το επίπεδο αριστείας επιστημονικής στα νέα κράτη-μέλη. Και για να συμπεράνω, ελπίζω ότι στον ορίζοντα δεν θα υπάρχει τέτοιο τόσο μεγάλο κενό όπως υπήρχε στα διαδοτικά. Η ε, κυρία Λόπες, ε, λέει ο πρόεδρος, είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε και καλά απόγευμα σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο Μόηδες για την παρουσία, την παρουσία του εδώ σήμερα. Η στήριξη στην έρευνα και τη γνώση είναι χωρίς καμία αμφιβολία μια, ένα αφήγημα επιτυχίας που συνεισέφερε στην ομαδοποίηση και την καλύτερη χρησιμοποίηση όλων των ε, γραμμών χρηματοδότησης στην Ευρώπη για τον τομέα αυτό. Όμως, ανησυχώ. Ανησυχώ πιο πολύ από ότι είμαι ικανοποιημένη για το μέλλον των έργων έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μου φαίνεται καθόλου σαφές Αυτή η έμφαση που δίνει η Κομισιόν ή στην ιδιωτικοποίηση των επενδύσεων ή στην έρευνα και ανάπτυξη είναι κυρίως το στοιχείο που με ανησυχεί περισσότερο. Δηλαδή η δημόσια πολιτική, η κρατική πολιτική ε, προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην συμπλήρωση των ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή έχουμε όλο και αυξανόμενο όγκο ιδιωτικών κονδυλίων με τον κίνδυνο να αφήσουμε στην άκρη τις περιοχές εκείνες όπου δεν προσφέρουν άμεση δυνατότητα κερδοφορίας και αντίστοιχα χρηματικής συνεισφοράς. Επομένως, διακρίνουμε μεταξύ των περιφερειών, εκείνων των περιφερειών που δεν έχουν επαρκώς παραγωγικό μοντέλο και τις ε, σύρουμε ή τις εγκλωβίζουμε όλο και περισσότερο στην τεχνολογική καθυστέρηση και αυτό οφείλεται στην χρήση των επενδυτικών ταμείων και ίσως θα χρειαζόμασταν εκεί καλύτερη συνέργεια με τα διαρθρωτικά και σε αυτό θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Ένα άλλος κίνδυνος είναι η αξιολόγηση της γνώσης να γίνεται μόνο όταν οδηγεί σε ιδιωτική κερδοφορία και όχι σε όφελος συνολικά για την κοινωνία ήταν, υπήρξε δυσάρεστη έκπληξη σε μένα για μία ακόμα φορά ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά από τον Επίτροπο ούτε στον κοινωνικό διάλογο ούτε στην ευρύτερη διαβούλευση ε, αλλά μιλούμε μόνο για ανάπτυξη βιομηχανική και επενδύσεων. Θα ήταν καλό να ενσωματώσουμε στοιχεία βελτίστων πρακτικών ή προϋποθέσεις κοινωνικής οικονομίας που θα μας οδηγούσαν σε θέσεις απασχόλησης υψηλότερης ποιοτητα συνολικά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Καρβεθόν Ρούις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ξεκινήσω και εγώ λέγοντα ότι μου φαίνεται μια έκθεση σαφώ ε, θετική. Μας δείχνουν τα στοιχεία, τα μεγέθη, την επιτυχία του προγράμματος. Και υπάρχουν και οι συστάσει στην ίδια την έκθεση τη Κομισιόν και αυτό που φαίνεται είναι ότι η Κομισιόν είναι ανοιχτή σε διάφορες συστάσεις που τις γίνονται και προχωρεί σε μία ανάλυση για τα όσα γίνονται στον τομέα της, ε, των επενδύσεων και της έρευνας. Τις συνέργειες μεταξύ των ταμείων ή την ανάπτυξη έργων ε, κοινή ωφελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όπως έλεγα και νωρίτερα πάντως, εγώ εμένα με ικανοποιούν ε, ιδιαίτερα τα μεγέθη που δείχνουν να φαίνονται από την έκθεση της Κομισιόν και επ' αυτού συγχαρητήρια. Επίσης είναι πολύ θετικό ότι το 1 ευρώ στην ε, επένδυση στην έρευνα δημιουργεί 11 ευρώ. 11 ευρώ ανταγωνιστικότητα συνολικών επενδύσεων ωφέλει στην οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζει το σύνολο της Κομισιόν και το Συμβουλίου έτσι, ώστε όταν ε, βρισκόμαστε σε αντίθετες περιπτώσεις ε, ε, εξοικονόμησης να μην εξοικονομούμε, να μην περικόπτουμε από προγράμματα τόσο πολύτιμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομίας της. Και βεβαίω είναι πάρα πολύ ουσιώδε να γνωρίζουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο του κάθε προγράμματο και του κάθε έργου είναι σημαντικό να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις κοινωνικές και οικονομικές, αλλά ε, είναι χρήσιμο να βλέπουμε και τι άλλες ωφέλειες ή κενά έχουν προκύψει από την προηγούμενη χρησιμοποίηση ή υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, αλλά και από τη διεθνή συνεργασία που έχει παρελά διδάγματα να μας δώσει για την πρόσβαση στην επιστήμη και στην ανοιχτή επιστήμη, είναι ε, χρήσιμο να μιλήσουμε για, μια, για την φάση των επενδύσεων, αλλά όταν μιλούμε για άδειες ευρυστεχνίας, αυτό δεν αφορά στον ίδιο βαθμό και δεν έχει τον ίδιο κοινωνικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς. Έχουμε τομείς όπως η υγεία, όπου οι άδειες ευρυστεχνίας θα ήταν καλό να γνωρίζουμε αν έχετε κάνει κάποια ανάλυση εσείς και πώς συνδυάζεται ε, ο αντίκτυπος επί των ιδιωτικών ε, επενδύσεων αλλά με το δημόσιο, με το κοινό συμφάρον. Σε πολλές από αυτές τις καινοτόμες νέες λύσεις ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η τελική τιμολόγηση, η πρόσβαση στην τελική ωφέλεια ή κερδοφορία πρέπει να διατηρούμε υπόψη μας λοιπόν τον αντίκτυπο, τον κοινωνικό αυτών των ωφελιών. Σας ευχαριστώ ρε Πρόεδρος, η κυρία Βίρκονεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο Μοέδας. Μια πολύ χρήσιμη παρουσίαση ως μέλη της Επιτροπής Ήτρε και πολλές από τις συστάσεις αυτές ε, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στα πλαίσια του προγράμματος ε, ορίζοντας 2020, εκπλήσωμε που είχαμε τόσο καλά αποτελέσματα στην αξιολόγηση πριν να γιατί τα σχόλια που εγώ είχα ακούσει σχετικά με το PP7 από τους ερευνητές και τις μικρές και μισές επιχειρήσεις ήταν ότι είχαμε τόσο ανεπτυγμένη γραφειοκρατία, τόσο περίπλοκους κανόνες που, τι να σας πω, εκπλήσωμε, που τα αποτελέσματα υπήρξαν τόσο θετικά. Βεβαίως υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών Γνωρίζουμε ότι η Ολλανδία είχε υποφεληθεί. Είχε υποφεληθεί επικυρίαρχα, θα μπορούσα να το πω έτσι, μεταξύ των άλλων χωρών, αλλά και εμείς, και εμείς στη Φιλανδία. Δεν μπορώ να πω. Ε, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον ότι η εικόνα του προγράμματος συνολικά, η φήμη του, είναι ότι είναι δύσκολο στην πρόσβαση. Και αξιολογώντας εμπειρίες των ενδιαφερομένων φορέων στη Φιλανδία, ε, ήταν έκπληξη που προέκυψε ότι μόνο το 10% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμμετείχαν στο 7. Μας είπαν ότι είχαν κάποιο πρόβλημα γραφειοκρατικής διαδικασίας. Ίσως να το περίμεναν ακόμη πιο δύσκολο και τελικά να τους φάνηκε πιο εύκολο το πράγμα στην πράξη. Εν πάση περιπτώσει, όπως γνωρίζουμε τώρα, αρκετά κρατημέλη καθότι έχουν οικονομικά προβλήματα, έχουν περικόψει τα κονδύλια έρευνα και ανάπτυξη και ήδη κατά τη διάρκεια του 7ου προγράμματο πλαίσιο ο ανταγωνισμό ήταν σκληρό και ξέρουμε ότι με τον ορίζοντα 2020 θα είναι ακόμη πιο σκληρό. Και πλέον αυτό που λένε οι ερευνητέ και οι ΜΜΕ είναι ότι έχουν έξοχα έργα και το πιστεύω, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί χρηματοδότηση πλέον γιατί υπάρχουν τόσε πολλέ υποβολέ και κάνουν τόση πολλή δουλειά προετοιμασία των υποβολών αυτών που ναι, εξαιρετικά είναι τα έργα, αλλά δεν μπορούμε να τα όλα. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να του βοηθήσουμε. Uh, thank you very much. Um, I may add very shortly, Mr. Mr. Commissioner. Uh... Αν uh, μου επιτρέπετε να προσθέσω σύντομα, κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος, εισήγαμε εμείς στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο κάποια απολύτως καινούργια σημεία. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα, μονολεκτικά ή δυνατόν, να μας αναφέρετε πέντε, ξέρω εγώ, καινούργιες ιδέες. Με μια βαθμολόγηση από 1 ως 10. 10 εξαιρετικά, ένα πολύ μέτρια. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερεύνηση. Πρώτη φορά που εισήχθη. Κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες Τρίτο σημείο. Έρευνα στι υποδομέ πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Τέσσερα. Ε, Εταιρικέ προκλήσει υπερεθνικέ. Και τέλος, Risk Sharing Finance Facility. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση αντιστάθμιση του κινδύνου που έχει και αντιστοιχήσει στο πρόγραμμα Juncker. Μία βαθμολόγηση εγώ θα ήθελα να μου κάνετε. Από το 1 στο 10. Γιατί αυτά ήταν τελείω καινούργια. 10 ε, επαναλαμβάνει το άριστα. Πολύ καλά. Θα ξεκινήσω με εσά, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, 10 δίνω στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο, Συμβούλιο. Όπου και να πάω στην Ευρώπη, όλοι μου λένε ότι καλύτερο του έχει συμβεί. Με τα κοινέ ε, τεχνολογικέ ε, πρωτοβουλίε θα έλεγα 9, επειδή το δεκάρι πάει στο ερευνητικό συμβούλιο. 9 λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικό και έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Ερευνητικέ υποδομέ. Θα έδινα ένα 8, γιατί νομίζω ότι μας έχει πάρει πολύ καιρό. Είναι εξαιρετική ιδέα, αλλά η υλοποίησή τη ε, καθυστερεί περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Κοινωνικές αλλαγές 10 είναι κρίσιμη σημασία σε αυτό το στοιχείο για την καινοτομία και την επιστήμη και μετά επιμερισμός των κινδύνων και σχετική διευκόλυνση και αυτή τη βαθμολόγω με 9 γιατί νομίζω ότι είναι ο σπόρος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έχουν ε, χρησιμοποιήσει αυτή την ιδέα της καινοτομίας. Εντάξει, σε όλα δέκα θα μπορούσα να δώσω. Απλώ ήθελα να σα ε, να δώσω, κάνω ιδιαίτερη μνήμα στο Ερευνητικό Συμβούλιο. Ήθελα να το βάλω στην κορυφή. Μετά, εν συντομία. Και να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ξεκινάω από τον κύριο Ρουβίκ. Μίλησατε για τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έκανε εξαιρετική δουλειά. 6,4 δις προς τις μικροπροσίες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος. Όμως πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Γιατί πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά της δημιουργίας της απασχόλησης για το μέλλον. Αυτή είναι το κύριο συστατικό και τη απάντηση προ ε, την Ευρωβουλευτή Μαρίζα Ματία ε, για την δημιουργία τη απασχόληση. Και μετά μιλήσατε για το εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει και να το βελτιώσουμε πολύ περισσότερο. Μετά. Ελπίζω να, ξέρω, να προφέρω καλά το όνομά σας, Μπάρμπαρα Κοντρίσκα, για ε, τους Προέδρους ERC. Ορίζον 2020 είχε 800 εκατομμύρια στο πρόγραμμα. Μέχρι τώρα, στα τέλη του 2015 δηλαδή, είχαμε περίπου 169 ε, συνδέσεις, 533 ε, ε, ε, συνεργασίες και 88 προεδρίες ΕΡΑ. Είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα Θα σας δώσω πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία της Πολωνίας. Αν θέλετε θα τα στείλω με mail. Μετά, η κυρία Λόπες. Καλό, καλό, σας απόγευμα. Ναι, ήθελα να σας αναφέρω. Es que hay que haber un equilibrio entre Υπάρχει ένα σαφή σχετισμό μεταξύ των ιδιωτικών και των δημοσίων πόρων για την ε, καινοτομία και για την επιστήμη. Το θεμελιώδε για την επιστήμη που οδηγεί σε νέα γνώση είναι ότι πρέπει να περνάει από δημοσίους πόρους και αυτό είναι ουσιώδες. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόγραμμα 2020 ορίζοντας πήγε σαφώ προ την κατεύθυνση αυτή. Διότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρεύνη ε, είχε ω στόχο να διατηρήσει αυτήν την ηγετική θέση που έχει η Ευρώπη για την ε, δημιουργία τη γνώση. Και για τη δημιουργία τη γνώση οι δημόσιοι πόροι, τα δημόσια κονδύλια είναι θεμελιώδης, θεμελιώδης σημασίας. Εγώ πάντοτε ήμουν υπέρ και πάντοτε επαναλάμβανα ότι το μεγάλο πλεονέκτημα μας στην Ευρώπη είναι ότι διατηρήσαμε τα δημόσια αυτά κονδύλια. Βεβαίως πρέπει να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι είναι πολύ σημαντικά να έχουμε και ιδιωτικούς πόρους που να μπορούν να συμπληρώνουν. Δεν είναι οι δημόσιοι πόροι που συμπληρώνουν αλλά στην ουσία και τα δύο είναι συμπληρωματικά. Και, τα, και αμφότερα είναι σημαντικά. Όταν δημιουργούμε νέα γνώση θα πρέπει μετά να την τροφοδοτήσω για τη δημιουργία νέων προϊόντων τα οποία τα δημιουργούν οι επιχειρήσεις. Ήθελα όμως να σας διαβάσω το μήνυμα αυτό και να σας βεβαιώσω ότι είμαι ένας από τους φονταμενταλιστές της διατομεακότητας της διαδικασίας αυτής της δημιουργίας νέας γνώσης και ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της όλης προσπάθειας. Δεν έχουμε καμία διαφορά δηλαδή σε αυτό. Για την κυρία Καβεθόν Ρούγες, να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκαιο. Θα έπρεπε να κοινοποιήσουμε πολύ καλύτερα το, την, την πολύ καλή απόδοση που έχουμε του 1 ευρώ προς τα 11 σε τελικό προϊόν, αλλά εγώ ήθελα να κάνω περισσότερα. Στο PP7 e ε, το 8% πήγαν σε ε, χώρες ε, συνδεδεμένες, το 85% περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο στους υπολείπους. Νομίζω ότι αυτό το σχετισμό θα έπρεπε να το βελτιώσουμε πάρα πολύ. Όσο δε για τις άδειε ευρυτεχνία ε, και τι εκκρεμότητε που έχουμε εκεί στον τομέα τη υγεία, δεν έχω, πρόσφατα τα, δεν έχω μπροστά μου τα... Και Τέλο. σα ευχαριστώ ε, για τα ερωτήματά σα. Ήταν ενδιαφέρον ο τρόπο με τον οποίο θέσατε το ερώτημα. Είπατε ότι πραγματικά έχω μείνει άναυδη από τα τόσο εξαιρετικά αποτελέσματα. Όμως νομίζω ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα έχουν πολλά μηνύματα και συμπεράσματα να μας ε, δώσουν. Για παράδειγμα, όταν μιλήσετε για την γραφειοκρατία, πράγματι ισχύει αυτό που λέτε και ο 2020 παρουσιάζει βελτιώσεις, αλλά πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Εξακολουθεί να υπάρχει γραφειοκρατία, το ακούω αυτό από πολλούς. Ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο κύμα απλούστευσης με σκοπό να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ταυτόχρονα όμω όλοι μου λένε ότι ο ορίζον 2020 είναι καλύτερο από πλευρά ε, περιορισμού τη γραφειοκρατία. Μετά είπατε κάτι το οποίο μου έχουν αναφέρει πέντες φορές, Η αντίληψη της δυσκολίας. Κάποιοι λένε, α, θα είναι πολύ γραφειοκρατικό θα είναι μεγάλη διαδικασία. Δεν μπαίνω καν στον κόπο να προσπαθήσω. Πρέπει να αλλάξουμε και την αντίληψη ε, στα κράτη-μέλη. Γιατί το πρόγραμμα Horizon 2020 είναι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο απλό. Όμως, σε ορισμένε χώρες υπάρχει ακόμα αυτή η αίσθηση ότι είναι δύσκολο, είναι επαχθέ. Και θα πρέπει αυτό να το αλλάξουμε. Και μου άρεσε αυτή η παρατήρησή σας. Γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να επαναπαυόμεθα. Πρέπει να το χαρούμε, αν θέλετε, να το γιορτάσουμε, γιατί αυτό δείχνει ότι αξιοποιούνται ε, στο έπακρον τα κονδύλια των Ευρωπαίων φορολογουμένων, αλλά δεν επαναπαυόμεθα, προχωρούμε γιατί πρέπει να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Πώς δηλαδή αυτή τη γνώση θα την ε, μεταφράσουμε σε καινοτομία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και την παρουσία σας εδώ σήμερα. Όπως είπατε και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για την πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστούμε που ε, θελήσατε και θέλετε και είστε διεθυμένος να έρχεστε στην Επιτροπή μας κάθε φορά που σας ε, προσκαλούμε. Thank you, dear colleagues. We go, we are... Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα περάσουμε στο σημείο 8, παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδική έκθεση σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ασφάλειας ε, της ενεργειακού ανεφοδιασμού, με τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς. Ο κύριος Βιν Όουεν είναι μαζί μας, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσίαση, ανταλλαγή απόψεων. Και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκπονήσει μια ειδική έκθεση για την ασφάλεια ενφοδιασμού και τη σύνδεσή της με την ε, ενιαία αγορά. Και έχει καταλήξει σε εννέα συστάσεις. Ε, πολύ σημαντικά όλα αυτά για μας. Ε, σας καλωσορίζουμε κύριε Βιμ Όουεν και θα μας παρουσιάσετε όλες αυτές τις ε, συστάσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για μας. Συστάσεις ε, που θα συνδιαμορφώσουν και τις εργασίες της Επιτροπής Ήτρε στο επόμενο διάστημα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λεγκτικού Συνεδρίου. Στα αριστερά μου είναι ο κύριος Έρκι Μούστ, επικεφαλής ε, της ομάδας. Και ο Γκάρεθ Ρόμπερτς, επικεφαλής του επιτελείου μου, είναι εδώ κοντά μας και του ευχαριστώ και τους δύο ε, για τα όσα έχουν κάνει για την έκθεση. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι έχω παρουσιάσει την έκθεση και σε αυτή την, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, την Επιτροπή Κοντ, την ε, προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχαμε κάνει μια πολύ καλή συζήτηση, με τα χαράς να ακούσω και τις δικές σας ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Περίπου 3,7 δις ευρώ έχουν καταναμηθεί από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεργικές υποδομές από το 2007 έως το 2013 και 7,4 δις, διπλάσιο δηλαδή ε, ποσό, προβλέπεται να χορηγηθεί μέχρι το 2020 στον ίδιο τομέα. Η ασφάλεια ενεφοδιασμού στην ενέργεια είναι κρίσιμη σημασία ζήτημα για την Ευρώπη ε, σε έναν ολένα και πιο αβέβαιο κόσμο. Για να το πετύχουμε πρέπει να ολοκληρώσουμε την ενιαία ενεργειακή αγορά και να μοιραστούμε την ενέργεια που ήδη διαθέτουμε. Όπως ξέρετε, η ενιαία αγορά ενέργειας είναι ε, το ρυθμιστικό ε, σύνολο υποδομών το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη ροή πέραν ε, των συνόρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο πρόσφατο νομοθετικό πακέτο, γνωστό και ως τρίτο πακέτο, υιοθετήθηκε το 2009 και το 2011. Το Συμβούλιο ανέφερε ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα το 2014. Ε, η δική μας ε, επιθεώρηση έχει ως στόχο να δει κατά πόσο η υλοποίηση των ε, αντίστοιχων μέτρων και οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών έχουν δώσει ακριβώς τέτοια ωφέλη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ενφοδιασμού. Καλύψαμε την χρηματοδότηση και τα μέτρα πολιτικής από το 2007 και μετά. Εξετάσαμε μελέτες περιπτώσεων σε τέσσερις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Εστονία, Λιθουανία και Σουηδία. από το λεγόμενο BIMIP, αυτή την περιοχή για το ε, σχέδιο διασύνδεσης που λέγεται BIMIP και τους, ε, τις περιοχές γύρω από τη Βουλγαρία, Πολωνία και Ισπανία. Εγώ προσωπικά επισκέφθηκα την Εστονία ένα πολύ καλό παράδειγμα, το λεγόμενο πρόγραμμα Estlink, στη Λιθουανία και στη Βουλγαρία πήγα επίση. Συμπεριλάβαμε 15 παραδείγματα συγκεκριμένων ε, προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο έλεγχό μα επικεντρώθηκε στην μετάδοση ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορά φυσικού αερίου μέσω ε, αγωγών και την αποθήκευσή του, ε, συμπεριλαμβανομένου και του LNG και τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα βασικά μα πορίσματα. Πρώτον, ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ολοκλήρωση τη ε, εσωτερική αγορά ενέργεια μέχρι το 2014 δεν επετέχθη. Παραμένουν προβλήματα ω προ την υλοποίηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Για παράδειγμα, οι ενεργειακέ ρυθμιστικέ αρχέ δεν είναι πάντα απολύτω ανεξάρτητε και ούτε πάντα έχουν όλε τι εξουσίε και του πόρου για να κάνουν σωστά τη δουλειά του σημαντικές διαφορές ε, μεταξύ των κρατών μελών στην οργάνωση ε, των αγορών ενέργειας μπορούν να αποτελούσουν τροχοπέδι για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Για παράδειγμα, ε, η διαδικασία για την προσδιορισμό των τεχνικών κανόνων, ούτως ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα στην αγορά ενέργειας, δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση. Υπάρχουν σημεία προόδου σε ό,τι αφορά την εμβαλωματική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις αγορές ενέργειας σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ε, τιμές χονδρικής της ενέργειας ε, στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό. Δεύτερον, οι ενεργειακέ υποδομέ δεν έχουν σχεδιαστεί για μια πλήρω ολοκληρωμένη αγορά. Οι υποδομέ σε ένα κράτο μέλο μπορούν να επηρεάσουν τι ενεργειακέ ροέ σε άλλο κράτο μέλο. Επομένω, κάθε χώρα πρέπει να είναι έτοιμη να αποτελέσει ε, χώρα διαμετακόμιση. Όμω, κάποια σημεία διασύνδεση δεν μπορούν να λειτουργούν σωστά, γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένα κεντρικά ε, κράτη-μέλη ε, ω προ τη διαμετακόμιση, όπω είναι η Γαλλία. Δεν υπάρχει γενικότερη αξιολόγηση αναγκών για να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες ω προ τι επενδύσει στι ενεργειακές υποδομές. Κάποιες από τις υφιστάμενε υποδομές δεν αξιοποιούνται στο έπακρον. Για παράδειγμα, στην Πολωνία έχουμε διασυνοριακές γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική ισχύ 5 ε, γιγαβάτ που δεν είναι διαθέσιμα για το εμπόριο εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ίδιες οι πολωνικές ε, αρχές, ο λόγωμενος TSO, για να αντιμετωπίσει ε, μη προγραμματισμένες ροές με τη Γερμανία. Η ανάπτυξη και πλήρης αξιοποίηση των υποδομών απαιτεί συνεργασία μεταξύ γειτονικών κρατών μελών. Επομένω, πρέπει να εξετάσουμε ε, τα, τα συστήματα αναμετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας σε και τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μετά, η οικονομική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στον τομέα αυτό έχει πολύ συγκεκριμένη συμβολή. Έχει διάφορα μέσα χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ε, δεν είναι ο βασικός στόχος η εσωτερική αγορά ενέργειας όπως έχουμε δει με συγκεκριμένα προγράμματα όπως το EPPR που δεν έχει επιτύχει ε, τον βασικό της στόχο που ήταν η οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, ε, επί των συστάσεων, μπορείτε να βρείτε βεβαίως και αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία και στην έκθεσή μας. Πρώτον, η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της ως προς την υλοποίηση του τρίτου πακέτου ενέργειας από τα κράτη-μέλη και ε, να κινήσει ειδικέ επί παραβάση όπου αυτό είναι απαραίτητο απέναντι στα κράτη-μέλη μέχρι τα τέλη του 2016. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους ρυθμιστικές αρχές είναι ανεξάρτητες, ε, έχουν επαρκείς πόρους και δεν περιορίζονται στο έργο τους. Η Επιτροπή επίσης οφείλει να διασφαλίσει ότι ο λεγόμενος ACER, ο Ευρωπαϊκός Φορέας ε, για, την για των ρυθμιστικών αρχών, έχει τις απαραίτητες εξουσίες και ομοδιότητες ε, για να κάνει το έργο του όπως πρέπει. Μετά, η Επιτροπή θα πρέπει να, να προαγάγει ε, τη διευρυμένη ανάπτυξη της, ενός ανεξάρτητου εμπορικού μηχανισμού. Θα πρέπει να αυξήσει τη διαδικασία Ε, της ε, θέσπισης ε, συγκεκριμένων διαδικασιών που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2015. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καθυστερήσεις ως προς την εσωτερική αγορά ενέργειας και πρέπει η ίδια η Επιτροπή να κατεβάσει τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις. Θα ήταν καλό να δούμε τι συμβαίνει και από αυτές τις καθυστερήσεις. Μετά, για την ηλεκτρική ενέργεια. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει ε, στόχους διασύνδεσης για την ηλεκτρική ενέργεια βάσει των αναγκών της αγοράς και όχι της ισχύω. Για το φυσικό αέριο θα πρέπει να επανεξετάσει η Κομισιόν ε, το μοντέλο ως προς την αγορά φυσικού αερίου και επειδή είναι αβέβαιη η αγορά και η ζήτηση, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν λύσεις λύσει προς την επέκταση ή ε, διαμόρφωση αγωγών φυσικού αερίου. Μετά, η Επιτροπή θα πρέπει να εντοπίσει ενεργειακές υποδομές που υφίστανται αλλά δεν αξιοποιούνται στο έπακρον και να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσει την πλήρη αξιοποίησή του ε, προ όφελο τη εσωτερική αγορά ενέργεια. Και θα πρέπει να διαρευνήσει τα ωφέλη από τη σύσταση περιφερειακών TSOs. Έβδομον, η Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει ε, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση επί των αναγκών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με γενικότερες προβλέψεις για το μέλλον είτε να τις εκπονήσει η ίδια είτε ο Acer. Γιατί έχει υποτιμήσει το παρελθόν, ας πούμε, τη ζήτηση φυσικού αερίου. Και τέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις ε, ως προς την υποβολή προτάσεων και αποφάσεων για την επιλογή συγκεκριμένων προγραμμάτων για χρηματοδότηση που υπόκειται στην κατάλληλη και εύρυθμη ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ε, με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή δέχτηκε τις περισσότερες από τις συστάσεις μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη θέση σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σαφή τα όσα είπατε και τα περισσότερα σχόλιά σας απευθύνονται στις χώρες μέλη, βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ώστε να χρησιμοποιήσει τι εξουσίε τη για να ασκήσει επιρροή μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τι χώρε μέλη. Στι χώρε μέλη, για να συνεργαστούν αυτέ και να δοθεί η δυνατότητα συνεργασία για να δημιουργηθεί η ενιαία αγορά ενέργειας. Τώρα, ε, αγαπητές και αγαπητοί, πρώτος Μπλάνκο Λόπε. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσάς κύριε εκπρόσωπε του Ελληνικού Συνεδρίου για τις πληροφορίες. Δύο ήταν οι παρατηρήσεις που κάνει η έκθεση και που μου φάνηκαν σημαντικές. Πρώτον, συμπεραίνεται ότι οι υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη δεν αρκούν, δεν είναι για μια πλήρη ενοποίηση της αγοράς. Τα διασυνδεμένα δίκτυα θα πρέπει λοιπόν να λάβουν μια πρώτη στην προτεραιότητα. Με δοθεί προτεραιότητα λοιπόν στα δίκτυα, γιατί αυτά είναι που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Εγώ διερωτώ Χρειάζεται να αποδείξουμε ακόμα περισσότερο με δεδομένα, με αξιολογήσεις και ούτω καθεξής για να διαπιστώσουμε ποια σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απομονωμένες νησίδες ενεργειακά. Αυτές οι ενεργειακές νησίδες δεν μπορούν να είναι συμβατές με μια ενιαία ενεργειακή αγορά. Όλοι μπορούμε να τις ε, εντοπίσουμε αυτές. Πότε θα τις απαντήψετε και με ποιες προσπάθειες ο Ευγένιος Τοσενόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το ότι κάνατε αυτού του είδους τον έλεγχο σε ένα τόσο σημαντικό τομέα για την ΕΕ. Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η έρευνα αυτή και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας. Πολλά λέτε στην εκθεσή σας, την οποία θεωρώ και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να μάθω από εσά σε ποιο βαθμό κατά την θεώρηση της καταστάσεως της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη που κάνετε εσείς. Πώς αξιολογείτε τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης αστάθειας. Δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης υπάρχουν εχμές της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, από την αιωλική ενέργεια. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν απειλή για άλλες χώρες. Μπορούν δηλαδή να οδηγήσουν σε μια αστάθεια της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχω μιλήσει μαζί του και στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού για ορισμένα οικονομικού χαρακτήρα θέματα. Και σήμερα όμως είναι σημαντικό να φτάσουμε μέχρι την ουσία των θεμάτων αντί να χρησιμοποιήσουμε συνθήματα και τίτλους. Τα νούμερα που έχουμε δείχνουν καθαρά ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπλοκη κατάσταση. Έχουμε καταβάλει προσπάθειες για να ολοκληρώσουμε την ενεργειακή αγορά τα τελευταία 6 χρόνια. Ωστόσο είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέτυχε στην προσπάθειά της αυτή να υπολογίσει δηλαδή σωστά τους στόχους της ενεργειακής στρατηγικής. Χωρίς όμως ορθούς υπολογισμούς είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι είδους υποδομές θα χρειαστούμε. Έχουν λοιπόν υπάρξει σφάλματα και στην επιλογή έργων και πολλά, πολλές χρηματοδοτήσεις χάθηκαν διότι κάποια από τα έργα αυτά σταμάτησαν στη μέση. Γνωρίζουμε ότι θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες το τρίτο ε, πακέτο. 19 χώρες μέλη σήμερα όμως δεν έχουν προχωρήσει τη μεταφορά αυτή. Ο κ. Όουεν αναφέρθηκε σε έναν αριθμό έργων. όταν μιλούμε για την περιοχή της Βαλτικής, όταν μιλούμε για την πολωνική στάση απέναντι σε ορισμένα από τα έργα. Ε, μου προκαλούν ησυχία και έκπληξη τα πράγματα αυτά. Το Ενεργειακό Συμβούλιο πρέπει να αναλύσει Όμως, ο οργανισμός ενέργειας δεν έχει την εξουσία να ζητήσει μέτρα από τις χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς αυτά δεν μπορεί, χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να προχωρήσει τη λύση αποφάσεων. Ευχαριστώ μεν το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να ρωτήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα τερματικά SGD. Μία από τις χώρες μέλη αποφάσισε να επενδύσει σε τέτοιους τερματικούς σταθμούς. Δεν βλέπω όμως άλλες χώρες μέλη να έχουν τη διάθεση να αγοράσουν το αέριο που θα βγαίνει από τους τερματικούς αυτούς σταθμούς. Χρειάζεται λοιπόν κάπως να ασχοληθούμε με την πραγματικότητα. Τον κύριο για την παρουσίαση. Ε, συμφωνούμε με τη θέση του ελεκτικού συνεδρίου και που καταγράφεται στην έκθεση πως για να πετύχουμε την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ιδιαίτερα της ε, ασφάλειας του ενεργειακού φοδιασμού είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια συνολική εκτίμηση των αναγκών που υπάρχουν σε υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση. Εξίσου είναι ορθή θέση που αναπτύσσεται στην έκθεση πω η ανάπτυξη των διασυνοριακών υποδομών απαιτεί την ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Εν τούτης, ο στόχο που τίθεται για ολοκλήρωση τη εσωτερική ε, ενεργειακή αγορά δεν πρέπει να παραγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να επιτελήσει το κράτο και δει ο κρατικό έλεγχο στη ρύθμιση τη ενεργειακή αγορά. Κατά νέα όψη μα για να μπορέσει να βελτιωθεί η ενεργειακή τροφοδοσία και να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια είναι απαραίτητο να υπάρχει και εθνική ευελιξία και να δοθεί ενισχυμένος ρόλος στις ε, εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Έκανε στην παρουσίαση του κύριο Σόμεν αναφορά ε, στις ε, επάρκεια των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Όμως κύριε Όεν, εσείς ποια μειονεκτήματα ε, θεωρείται ότι υπάρχουν στη μεταφορά του ελέγχου της ενεργειακής αγοράς σε κοινοτικό πλαίσιων πάνω από τα εθνικά ρυθμιστικά προγράμματα. Ε, δυστυχώς επίσης η έκθεση εξέτασε περισσότερο τις περιπτώσεις έξι κρατών μελών. Ωστόσο θα ήταν σημαντικό να έχουμε μια λεπτομερή εικόνα από το ελεκτικό συνέδριο της σημερινής κατάστασης και των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει προγραμματισμός για την εξέταση των περιπτώσεων και άλλων κρατών μελών. Και να φέρω ένα παράδειγμα, ε, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η περίπτωση της Κύπρου, που όπως επισημαίνεται στην έκθεση, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ενεργειακής νησίδας. Είναι ένα κράτος δηλαδή απομονωμένο από τα ενεργειακά δίκτυα. Εν τούτης βεβαίως με την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών και τη στήριξη τη αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που διαθέτει μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο και για την εσωτερική ενεργειακή τροφοδοσία αλλά και για την ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια τη Ένωση. Επίση, στην Κύπρο μπορεί να εφαρμοστεί με πολλά ωφέλη και πρόταση παραψήσεται στα συμπεράσματα για δημιουργία τερματικού σταθμού υγροποίηση φυσικού αερίου ω μια εναλλακτική πρόταση στην εκτεταμένη κατασκευή αγωγό φυσικού αερίου ε, μάλιστα αξιοποιώντα και τα κοιτάσματα τη ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική μετεξογείου που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, thank Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόφοντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω για την ε, εξαιρετική έκθεση και τις πολύ χρήσιμες συστάσεις και συμπεράσματα. Συμφωνώ με τους συναδελφούς λέγοντας ότι μέχρι στιγμής η εσωτερική ενεργειακή αγορά δεν λειτουργεί και θα χρειαστούμε ένα μεγάλο βήμα για να το επιτύχουμε αυτό. Μου άρεσαν τα συγκεκριμένα παραδείγματά σας σχετικά με το πού υπάρχουν οι ελλείψεις, τα προβλήματα, αυτό που είπατε για τη Γαλλία και άλλες χώρες. Μήπως μπορείτε να επιταθείτε περαιτέρω, γιατί χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα από τα παραδείγματα. Επίσης αναφερθήκατε στην σύσταση παριθμών 2, για παράδειγμα. Την ε, έκθεση της ΕΙΣΑ για την παρακολούθηση της αγοράς. Δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Και δυσκολεύονται να, να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά από τα κράτη-μέλη. Σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς ότι το ζήτημα για την ΕΙΣΑ της εντολής τους αλλά και τους πόρους, των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους ε, είναι πολύ σημαντικό ε, Ω προ το διάλογο και τη συνεργασία που έχουν και με την Κομισιόν. Επίση σε αυτά τα σημεία ε, κυκλοφοριακού προβλήματο που δημιουργούνται. Είναι και αυτό ένα ζήτημα για την εσωτερική ενεργειακή αγορά και δεν ξέρω αν το έχετε δει και αυτό. Για τους δε νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή σύσταση αλλά είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να παραδοθεί βραχυπρόθεσμα. Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την πρότασή σας για το πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τη σύσταση αυτή. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Προφανώς υπάρχουν και διαδικασίες ε, κύρωσης, για να μην αναφερθούμε στο δικαστήριο. Παραμάνων ως τελευταίο βήμα. θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπόρχαρτ, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Ενιακή Αγορά, τι προτάσεις έχετε από πλευρά σας. Και τι κάνετε για να ενθαρρύνετε τα, τα κράτη-μέλη για να πάνε προς την ιστορική ενέργεια αγορά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Όουεν και την ομάδα του για την έκθεση αυτή. Ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό μοιραζόμαστε τα πορίσματα και τα συμπεράσματα και ε, το ίδιο ισχύει και για τις συστάσεις. Τώρα, αυτό που πρέπει να υπογραμμίσω είναι ότι πολλά από αυτά που συστήνονται και πολύ σωστά υπογραμμίζονται από την έκθεση έχουν ήδη δρομολογηθεί από την Κομισιόν. Και αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξη. Εδώ χάνουμε το μικρόφωνο του ομιλητή. Ε, είναι χρήσιμο λοιπόν να υπογραμμίσουμε και κάποια σημεία που ανέφεραν και κάποια μέλη της Επιτροπής. Να ξεκινήσω την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ναι, δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν είμαστε εκεί που έπρεπε. Το 2014 ήταν μια προθεσμιακή ημερομηνία, αλλά πρέπει να δούμε προς το μέλλον για να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε τα απαραίτητα ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την εσωτερική ενεργειακή αγορά το συντομότερο δυνατό. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εκφράζει και η έκθεση και κάποια μέλη της Επιτροπής ότι δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα, όλα τα κράτη-μέλη θα, θα συμμορφούνται προς το τρίτο ενεργειακό πακέτο και εδώ μπορώ να σας πω ότι το φθινόπωρο πέρυσι ολοκληρώσαμε τις τελευταίες εξετάσεις συνειακές νομοθεσίες όλων των κρατών μελών, όλων, και τουλάχιστον για την τρίτη δέσμη έχουμε ήδη εκκινήσει όλες τις διαδικασίες παράβασης που απαιτούνται. Βεβαίως βρισκόμαστε σε διαφορετικές φάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε γνωμοδότηση, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε οδηγηθεί ήδη στο δικαστήριο, σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε σε πρώτη ειδοποίηση κτλ. και εκεί που έχουμε ολοκληρώσει την παρακολούθηση είμαστε στην πιλωτική επιστολή. Αυτή τη στιγμή διερχόμεθα δηλαδή τη διαδικασία στις διάφορες αυτές φάσεις. Για τους κώδικες δικτύου, και εδώ με λυπεί κάπως το γεγονό ότι μεταφέρεται τόσο ευκριτικά το θέμα αυτό, διότι η κατάσταση σήμερα δεν είναι και τόσο κακή. Στο φυσικό αέριο, οι 4 εκ των 5 κώδικες έχουν υλοποιηθεί, λείπει ο κώδικας για τα τέλη, ο οποίος θα δοθεί στην Επιτροπολογία το Μάρτιο, στην ηλεκτρική ενέργεια. Ε, κινούμαστε προς 9 κώδικες, εκ των οποίων τέσσερις έχουν ολοκληρωθεί στην Επιτροπολογία, τρεις έχουν συγχωνευτεί σε έναν και θα μεταφερθούν τον ερχόμενο μήνα στην Επιτροπολογία, δύο απομένουν και μου ζητήθηκε να επεξεργαστούμε τι κάνουμε με αυτούς και γιατί τους έχουμε κρατήσει πίσω. Είναι πράγματι ένας από αυτούς ο κώδικας ε, εξορρόπησης, ε, πολύ σημαντικός για την ηλεκτρική αγωνά και για την προσέλευση εναλλακτικών πηγών στην αγορά, όπως και ο κώδικας ανάκτησης Restoration Code. Ε, εδώ όπως γνωρίζετε ίσως προετοιμάζουμε νομοθετικές προτάσεις για το νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παραλλήλως νέα νομοθεσία για την ε, ετοιμότητα έναντι κινδύνων για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι δύο αυτοί κώδικες ενέχονται στενά, συνδέονται στενά και πρέπει σε πρώτη φάση να δούμε τι πρέπει να πάει στην νομοθεσία και τι πρέπει να μείνει στις κώδικες. Αυτή η δουλειά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εδώ είναι η τελική μου απάντηση. Δεν θα περιμένουμε τη δουλειά αυτή μέχρι ότου να είναι έτοιμη οι νομοθετικές προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε και θα έρθουμε στην επιτροπολογία στο πρώτο εξάμεινο του έτους. Εντός του πρώτου εξαμήνου. Απλώς ξεκαθαρίζουμε πλέον σε, τελική, τελικό στάδιο τι πρέπει να πάει στην ομοθεσία. Και προχωρούμε κανονικά. Συνολικά λοιπόν πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο κακά τα πράγματα. Υπό αυτήν την έννοια. Και πολλά από αυτά που προκύπτουν ως στάσεις από πλευρά σα έχουν ήδη γίνει. Για τις υποδομές, το να λέμε ότι δεν υπάρχει συνολική αξιολόγηση των αναγκών, είναι κάπως υπερβολικό κάτι την άποψή μου. Είχαμε 10 χρόνια σχέδια ανάπτυξης ε, δικτύου, ε, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα. Από εκεί πέρα βεβαίως συμφωνώ με την ε, έκθεση του συνεδρίου και αυτή που αναφέρθηκε εδώ, ότι πρέπει να δούμε και τους αριθμούς των PCI. Και εδώ το σκεφτικό είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο το 2017 για να ανοίξουμε τον κανονισμό 10E του χρόνου και να καθορίσουμε εκείνα τα PCI που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ιστορικής αγοράς ενέργειας. Μετά σε δεύτερη κατηγορία θα είχαμε τα υπόλοιπα PCI και σε τρίτη κατηγορία θα ήταν τα έργα εκείνα που είναι σε μεθοριακές περιοχές με γειτονικές χώρες και εδώ μιλούμε για την ε, εκεί κοινότητα. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απολύτως τις υποδομές τις διασυνοριακές. Βεβαίως, εδώ έχετε απόλυτο δίκαιο. Και αναφερόμαστε στις αντίστροφες ροές. Είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό με τις μακαροπρόθεσμες συμβάσεις. Η στόχευση της λεκτικής ενέργειας, το κάνουμε αυτό. Βλέπω ότι μου δείχνετε ότι πρέπει να επιταχύνω, λέει ο μιλητής, για τις στρατηγικές υποδομές. Και μερικοί αναφέρονται και στο υγραέριο. Υπάρχει στρατηγικό έγγραφο 10 Φεβρουαρίου που θα βγει και εδώ έχουμε 9 συγκεκριμένα μέτρα υποδομών για το αέριο ώστε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την, ε, τη χρησιμοποίηση του LNG. Περισσότερη ισχύ σε αρμοδιότητα για την ASA. Βεβαίως και θα δείτε μέχρι το τέλος του έτους την ομοθετική μας πρόταση για τις πρωτοβουλίες ενεργειακού σχεδιασμού όπου θα δώσουμε περισσότερες εντολές στην ΕΙΣΑ και θα εξασφαλίσουμε ότι θα έχει άμεση πρόσβαση σε απαραίτητες λεωφορείες. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι με τα κράτη-μέλη, αλλά με τους διανομής. Έχουμε τους περιφερειακούς διανομής και συμφωνώ με το μέλος που, που είπε ότι αυτό θα έρθει μετά. Βεβαίως η αγορά θα το φέρει, δεν πρέπει να το επιβάλλουμε, αλλά θα επιμείνουμε εξ αρχής στην περιφερειακή συνεργασία μεταξύ μεταξύ διανομέων και θα δημιουργήσουμε δίκτυα εκεί που θα πρέπει να συνεργαστούν. Οι διαχειριστές δικτύου. Τώρα, δεν πρέπει να υπάρχει επίσης προκαθορισμένη χρηματοδότηση έργου που σχετίζεται με κράτος μέλος του οποίου η ενεργειακή αγορά δεν συμμορφούνται προ την τρίτη δέσμη. Ξαναχάνουμε το μικρόφωνο του μιλητή. Τώρα, έχουμε, επειδή τα, οι του ΣΕΦ δεν, δεν απονέμονται στα κράτη-μέλη, αλλά σε ιδιωτικέ επιχειρήσεις και TSOs. Και θεωρούμε ότι οι συνολικές προποθέσει θα τιμωρούσαν τις επιχειρήσει και τους διαχειριστές δικτύου που δεν είναι υπεύθυνοι για την τρίτη δέσμη και θα καθυστερούσε αρκετά πολλά σημαντικά έργα. Είχα όμως μια ή ε, κάπως άτυπη συζήτηση με τον κύριο, Σο, με τον κύριο Ον και μου έδωσε ε, καλές ιδέες. Αυτό που πρέπει σήμερα να τοποθετήσουμε δεν είναι μια συνολική, ένα συνολικό πλαίσιο προϋποθέσεων, αλλά σε σχέση με τα έργα να έχουμε ένα κριτήριο το οποίο να συνδέεται με τον διασυνοριακό αντίκτυπο. Αυτό θα μπορούσα να το προεκτείνω μάλιστα λέγοντας ότι εντός του κριτηρίου θα πρέπει να δούμε και το κατά πόσον στα συνδεδεμένα κράτη-μέλη γίνονται σεβαστοί οι κανόνες αγοράς κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζουν την πλήρη χρησιμοποίηση και αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου στοιχείου υποδομή. Και αυτό ενσωματώνεται στην αξιολόγηση. Και σας δίνω παράδειγμα. Θα έδινα 0 από 5, γιατί αυτή την κλίμακα χρησιμοποιούμε, αν σε κράτος μέλος είχαμε απαγόρευση εξαγωγής. Διότι αυτό θα κατέστρεφε απολύτως την χρησιμότητα Τη συγκεκριμένη υποδομή. Εάν το δικαστήριο ε, προτιμήσει να το κάνει στοχευμένα ε, εκτός, εντός διαδικασίας της στοχευμένης ε, της αξιολόγησης ΣΕΦ τότε θα μπορούσε να αποδεχθεί και την ένατη σύσταση που ήταν η μόνη που δεν είχε δεχθεί. Και ε, δύο σχόλια για αυτά που ακούστηκαν από τα μέλη η ενεργειακή είναι η προτεραιότητα που πρέπει να φτάσει στο τέλος της. Ρητή προτεραιότητα για την χρηματοδότηση της ΕΦ. Ε, να ανακοινώσω ότι εδώ έχουμε ήδη δύο επιτυχίες. Την διασύνδεση Πολωνίας-Λιθουανίας εκεί τελειώσαμε με την ενεργειακή νησίδα Βαλτικές. Και το δεύτερο βήμα Εστονία, Βιλανδία θα ολοκληρώσουμε και με την κατάσταση φυσικού αερίου ενεργής νησίδος ε, Φιλανδίας. Δηλαδή, εκεί έχουμε διοχετεύσει τους πόρους ΕΦ και ήταν ένα από τα σημεία συμφόρησης που είχαν αναφερθεί. Ο κύριος ε, Χομπονόφσκι αναφέρθηκε στα loop flows που μπορούν να είναι επιζήμια για άλλα δίκτυα. Αλλά και στην πρωτοβουλία ενεργειακού συνδυασμού θα ασχοληθούμε και με την τιμολόγηση. Και νομίζω ότι με αυτά ελπίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Μας φάνηκε πάρα πολύ σαφές αυτό που είπατε. Τώρα, έχω να σας ρωτήσω, κύριε Όουεν, μάλλον αν θέλετε πρώτα να σχολιάσετε ή να δώσετε κάποιες συμβουλές, προς τα πού να κατευθυνθούμε από εδώ και μπρος, ως ελεκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη σας, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποδοχή που επιφυλάξατε στην έκθεση. Θα απαντήσω σύντομα στα μέλη της Επιτροπής σας που έθεσαν ε, ερωτήσεις που έκαναν σχόλια και θα κάνω μια σύντομη, ε, ένα σύντομο σχολιασμό των απαντήσεων της Επιτροπής. Πλάνκο Λόπες μίλησε για μείωση επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό είναι ότι η διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι σχετικά μικρό μέρος της χρηματοδότησης της αγοράς. περίπου 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ενώ δίνει 14 δισεκατομμύρια ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το TSO. Είναι μικρό μεν, μεν μέρος της χρηματοδότησης, είναι όμως ένα μήνυμα διότι είναι τα ε, χρήματα του φορολογουμένου τα οποία διαθέτει στην επένδυση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, είναι σωστό οι επενδυτικέ αποφάσει να λαμβάνονται με σωστό τρόπο στο επίπεδο ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Να αποδώσει το δυνατόν περισσότερο κάθε ευρώ που δαπανάται σε τέτοιες επενδύσεις ώστε να γίνονται επενδύσεις σε σωστά έργα. Το Κενόσκι. Μιλήσατε για αυστηρά σε ό,τι αφορά την παρουσίασή μου. Δεν είναι βέβαια η πρόθεση μου αυτή. Όμως δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου είναι να τα πούμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε βασισμένα στις ενδείξεις και στα δεδομένα. Και νομίζω ότι όντως έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο μέχρι να φτάσουμε στην πλήρη υλοποίηση της ε, ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Ρωτήσατε τώρα και σχετικά με κίνδυνο αστάθειας και ε, την, ε, τα πίκα αυτά τις εχμές αυτές της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την γερμανική ολική ενέργεια. Είναι γεγονό ότι είναι σημαντική πρόκληση οι εχμές αυτές μέσα στα ηλεκτρικά δίκτυα. Μεγάλη πρόκληση για όλους τους μετέχοντες. Μια ενιαία ενεργειακή αγορά σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο είναι καταρχήν καλή ιδέα, διότι διαφοροποιεί τον κίνδυνο. Μπορεί να φυσάει ο αέρας κάπου, αλλά να μην φυσάει αλλού. Μπορεί να λάβει ο ήλιος κάπου ενώ αλλού να είναι σκοτεινά. Έτσι, μέσα στα πλαίσια ενός ε, τέτοιου ε, δικτύου διαφοροποιείται ο κίνδυνος και γι' αυτό είναι καλή ιδέα η ενιαία ενεργειακή αγορά και ιδίω στο πολωνογερμανικό πλαίσιο θα βοηθήσει μια ρύθμιση TSO ε, και η μεγαλύτερη διάθεση στο εμπόριο αυτών των εχμών ε, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο από τη Γερμανία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στην Πολωνία και να αντιμετωπιστούν έτσι κάποια απρόβλεπτα. Κύριε Μπαλτσίτη, σε ευχαριστώ για τις παρατηρήσει σα. Με ακούσατε δύο φορές. Ελπίζω ότι βεβαίως η παράληψη είναι η, η μετά Ελπίζω να σα βοήθησε αυτό. στην παράγωγο 31 της εκθέσεώς μας και επανέρχομαι και σε κάτι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι έχουμε 10 χώρες μέλη τα οποία είναι αντικείμενο διαδικασιών παραβιάσεως και έχουμε και άλλα 15 μέλη στην διαδικασία διαλόγου που ακολουθεί την κίνηση αυτή και ορισμένες ακόμη που θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα λάβουν επιστολή ή όχι. Υπάρχει, υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που παρακολουθεί τις υποθέσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι θα δώσει στον, στην ΑΣΕΑ τις εξουσίες που οφείλει να διαθέτει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και μιλούμε για νέες εξουσίες. Εμείς δεν πήγαμε μέχρι εκεί, αντιλαμβάνομαι όμως την αξία του επιχειρήματος υπέρ της ιδέας αυτής και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον για την ΕΣΑ. Ο κύριος Σιλικιώτης ρώτησε σχετικά με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Νομίζω ότι προσφέρουμε στην έκθεσή μας επαρκείς ενδείξεις για το αν είναι ανεξάρτητες ή όχι και εάν είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενες ή όχι και αν συμμετέχουν όσο θα έπρεπε στις συζητήσεις της ΕΣΑ. Και θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά μαθαίνουν οι χώρε μέλη από τα λάθη και από τι καλύτερε πρακτικέ που εφαρμόζουν. Με ρωτήσατε επίσης για το εάν μπορώ να πω περισσότερα για άλλε χώρε μέλη. ο ίδιος ο Σιλικιώτη μίλησε ιδιαίτερα για την Κύπρο. Βέβαια δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε μια έκθεση. Είναι πολύ ευρύ το πεδίο. Εγώ είμαι αρμόδιο πάρεδρος και για δύο εκθέσει που θα έρθουν του χρόνου και ε, θα έχουν σχέση με τις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής σας. Συζητούμε για αυτή την δαπάνηση ενός ευρώ ανά πέντε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματικούς στόχους και για χώρες όπως η Λιθουανία. Αλλά για να απαντήσω στον ε, κύριο Σιλικιώτη, είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια το θέμα που έθεξε για το δυναμικό της Κύπρου. Ε, προ δύο εβδομάδων ανακοινώσαμε το πρόγραμμά μας για το 2016 και είπαμε ότι η ενέργεια και κλίμα είναι μείζον θέμα για μας στο πρόγραμμα εργασιών μας του 2016. Και βεβαίως απηχεί αυτό την σημασία του θέματος στον ε, ορίζοντα 2020. Και θα επανεξετάσουμε ενέργεια και κλίμα υπό δική μου ευθύνη ε, μέχρι την ε, άνοιξη του χρόνου. Και στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσω και τα κυπριακά θέματα που έθεσε ο Σιλικιώτης γιατί βέβαια ε, οι νησιωτικά κράτη είναι σημαντικά από την άποψη αυτή. Κύριε Κόφωτ, ζητήσατε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε βάλει τέτοια πολλά στο κείμενο της εκθέσεώς μας. Έχουμε μάλιστα και ε, αντίτυπα σε χαρτί, που βεβαίως κάτι τέτοιο ε, το αποθαρρύνει το κοινοβολείο, που είναι paperless όπως γνωρίζετε. Ε, πολύ ευχαρίστω να τα λάβετε όμως και αν θέλετε με τον συνεργάτη μου μπορείτε να μιλήσετε για πιο ειδικά θέματα και για τα project για τις περιοχές που εξετάσαμε. Να πω λίγα λόγια για το ποιοι είναι οι τομείς που έχουν το υψηλότερο δυναμικό σε ό,τι αφορά να γίνουν χώρες διαμετακομιδής και εποφελία των δικών τους καταναλωτών αλλά και ε, των άλλων. Χωρίς να ασκώ καμία κριτική, έχω σημειώσει δύο χώρες. Η Γαλλία ενδεχομένως είναι μια πολύ σημαντική χώρα transit και για το αέριο και για το ηλεκτρικό ρεύμα, αν και υπάρχουν περιορισμοί μέσα στην ίδια την γαλλική εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά ε, τον όγκο ρεύματο που μπορεί να ε, διοχετεύσει, αλλά το ίδιο και η Πολωνία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους interconnectors που υπάρχουν μέσα στην ίδια την Πολωνία και κυρίω στο βορειοανατολικό μέρο τη. Πολύ ευχαρίστω να επεκταθούμε σε αυτό εφόσον επιθυμεί κάποιο. Δεν είναι λοιπόν μόνο ζωτική σημασία τα διαμεθοριακά ε, σχέδια και διαμεθοριακά ε, έργα. Πολλά από τα PCI τη είναι και αυτά που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση αχμών μέσα στις ίδιες τις χώρες. Τώρα, Πάλι και εδώ και σε άλλα θα έβαζα τις βέλτιστες πρακτικές Σουηδία και Δανία για παράδειγμα. Όπως και το Έσλιν 2, ο σταθμός δηλαδή των Φιλανδών και Εστονών, τη συνεργασία για τον σταθμό αυτό. Μιλήσατε κύριε Πρόεδρε και εσείς για διαδικασίες προσφυγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε όμως. Ευχαριστώ τον κύριο Μπολκχατ για τις ε, εγγύησεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρχικά τα έχει απορρίψει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που τα επανείδε. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρός σας, ο Επίτροπος Σεφκοβιτς, ξεκαθάρισε μιλώντα για το Nord Stream 2, νομίζω όμω ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και ευρύτερα. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει έργα υποδομή μόνον εφόσον αυτά είναι συμβατά με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Και χαίρομαι που οι αξιωματούχοι του επιμένουν στην ε, τήρηση των όρων αυτών. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρασχολιασμό των όσων βλέπουμε. Ευχαριστώ λοιπόν για τις ερωτήσεις σας και ελπίζω με τις απαντήσεις μου να σας ικανοποίησα. Ευχαριστώ. Προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος τα λεγόμενα PCIs, γιατί κάποιες φορές είναι ασαφές. Προγράμματα κοινού ενδιαφέροντο, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό τομέα. Σα ευχαριστούμε πολύ όλους για αυτή την πολύ καλή συζήτηση για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και την έκθεση του ελληνικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Uh, well, next point, nine. Το number nine. Στο σημείο 9 τώρα. Μελέτη σε ό,τι αφορά την αγορά σε σχέση με το διάστημα. Λόρα Ντελπόντ είναι η καλεσμένη μας από το Κέντρο Βιομηχανικών Ερευνών. Επιθυμία μας ήταν ε, να έχουμε ένα τύπο προσκεκλημένο. Το στείλαμε στο Τμήμα Πολιτικής ως ε, Επιτροπή Ήτρε. Αυτή η μελέτη λοιπόν που έγινε από το Τμήμα Πολιτικής ε, εκ μέρους της ε, Επιτροπής Ήτρε έχει ως στόχο Space Market Update. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, ζήτηση για δεδομένα, διαστημικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η διαστημική πολιτική είναι το μέλλον. Ιδίως αυτά που σχετίζονται με τα προγράμματα Κοπέρνικος και Γαλιλαίος. Τα ευρωπαϊκά διεθνικά προγράμματα, στα οποία έχουμε δαπανίσει πολλούς πόρους και σίγουρα θα δαπανίσουμε και άλλους στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αξιοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχουν. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε τα στοιχεία σας την έκθεσή σα. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Με τα χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα να σας παρουσιάσω τα ευρήματα αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ε, έκθεσης σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των διαστημικών τεχνολογιών στις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γιατί θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη και σημαντική αυτή η έκθεση για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει σχεδόν 6 δις ευρώ για να ε, οικοδομήσει τις δικές της διαστημικές υποδομές και στην ε, σημερινή κατάσταση βλέπουμε ότι 11 δι έχουν ε, τεθεί κατά μέρο ακριβώ για αυτές τις ανάγκες. Πρέπει λοιπόν, ε, βλέπουμε ότι πρέπει να δώσουμε αυτόνομες και ανεξάρτητες ε, διαστημικές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον γιατί η ανάπτυξη δορυφορικών βασικών υπηρεσιών και προϊόντων σίγουρα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και στρατηγικής. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξουν ε, κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Αυτό αποτελεί μια ε, στρατηγική πρόκληση ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ο στόχο και αυτή της μελέτη, Να δούμε ποιε είναι οι πιθανές κατευθύνσεις μπορεί να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαστημικών δεδομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για να εκπονήσουμε αυτή τη μελέτη, συνδυάσαμε διαφορετικές πηγές δεδομένων, κάναμε μία ανάλυση ε, ελέγχων βάσει ε, μελέτης, μελετών περιπτώσεων, αναθεώρηση εγγράφων πολιτικής και κανονισμών. Ταυτόχρονα όμως, εντάξαμε και αυτή την ανάλυση εγγράφων ε, συνδυάσαμε με διαφορετικές κατηγορίες εφαρμένων μερών, συμπεριλαμβανομένων και των τελικών χρηστών. Και πρέπει να πω ότι είμαστε ιδιαίτερω ευγνώμονε προ όλου όσοι συνέβαλαν στη μελέτη αυτή με την ε, γνώση και εμπειρογνωμοσύνη τους, γιατί μας έδωσαν πολύ σημαντικά στοιχεία. Ποια είναι λοιπόν ε, ποιε είναι οι ευρωπαϊκέ επενδύσει. Υπάρχουν ναι, δύο βασικά προγράμματα ναυαρχίδε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γαλιλαίο και το Κοπέρνικο. Το Γαλιλαίο είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ε, δορυφορική πλοήγηση. Είναι το αντίστοιχο τεσσοδύναμο του αμερικανικού GPS, αλλά έχει αναπτυχθεί καθαρά και μόνο εκτός στρατιωτικού πλαισίου βελτιώνει την ακρίβεια και αξιοπιστία του GPS και ήδη είναι λειτουργικό το Γαλιλαίο. Αποτελείται από ένα σύνολο 30 δορυφόρων και επιδάφιων ε, υποδομών. Το Κοπέρνικο θέλω είναι διαφορετικό. Είναι ένα σύστημα ε, γεωπαρατήρησης. Μας επιτρέπει δηλαδή να παρατηρούμε τη γη από το διάστημα και μας έχει δυνατότητα να δίνουμε χωροταξικές ε, πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη δημόσια πολιτική, σε πολλούς τομείς όπως είναι η ατμόσφαιρα, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια πολιτών και το καθεξής. Όλα και τα δύο αυτά προγράμματα είναι σε διαφορετικά στάδια της ε, διαδικασίας τους, ε, αναμένεται να προωθούμε στο 2020. Όταν εξετάζουμε Τώρα την κατάντη διαστημική αγορά έχουμε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμογές ε, σε μία σειρά δημοσίων και ιδιωτικών χρηστών. Αυτές οι επιχειρήσεις ε, γενικά δεν συνδέονται με την παραδοσιακή διαστημική αγορά, όμως βασίζονται ε, στην διαστημική αγορά για την παροχή δορυφορικού σήματος στην περίπτωση των εφαρμογών που απορρέουν από το Γαλιλαίος ή εικόνες, διαστημικές εικόνες στην περίπτωση του Κοπέρνικος. Πώς έχει κατάσταση στην αγορά. για τα δύο αυτά προγράμματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι δύο αγορές ανοίγουν, μεγαλώνουν και υπάρχει κυριαρχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως ό,τι αφορά την παροχή ε, υπηρεσιών που επιφέρουν τη αξία. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με τις ΗΠΑ Πολιτείες, η αύξηση των διαστημικών υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερη από αυτό που αναμέναμε. Και αυτό οφείλεται κατά βάση στο παρελθόν ότι η Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη και καταγερματισμένη αγορά. Η Ευρώπη λοιπόν χρειάζεται ε, κάποιους ε, παράγοντες προσέλκυσης ε, που θα επιτρέψουν ε, τις επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Οι δύο αγορές έχουν ε, ειδικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση του πρώτου προγράμματος ήδη έχει αναπτυχθεί Ξέρετε, ας πούμε, ήδη το σύστημα πλοήγησης μέσα στα αυτοκίνητα. χάρη στην ε, μεγάλη διείστηση των ε, smartphones ε, και τη οικονομία των εφαρμογών έχει ήδη αναπτυχθεί ιδιαίτερο. Δύο σημαντικοί παράγοντε ανάπτυξη των εφαρμογών που βασίζονται από το Γαλιλαίο είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων και τα αυτόνομα οχήματα. Στην περίπτωση της αγοράς παρατήρησης της γης είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα γιατί είναι αναδυόμενη η αγορά αυτή. Αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά αλλάζει πολύ γρήγορα για να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, στην αγορά κυριαρχούν ε, δημόσιοι και θεσμικοί επενδυτές και πελάτες, ενώ οι νέες υπηρεσίες ε, αναπτύσσονται περισσότερο για τις αγορές νης. Βλέπουμε λοιπόν δύο τομείς που έχουν υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης γεωργία και η No Life Insurance. Άλλος κινητήριο μοχλό ανάπτυξης μπορεί να είναι η πώληση γεωχροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό με, την, με τις υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης. Εξετάσαμε και τους περιορισμούς στη χρήση δορυφορικών δεδομένων στην Ευρώπη. Έχουμε ταξινομήσει σε πέντε κατηγορίε αυτέ του περιορισμού. Ε, περιορισμού πολιτική, αγορά, διακυβέρνηση, τεχνικών ζητημάτων και έλλειψη ε, προσόντων και δεξιοτήτων. Τα έχουμε ταξινομήσει με βάση ε, διάφορου βαθμού κρισιμότητα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, θα ήθελα να αναφέρω αυτά που έχουμε εντοπίσει ως κοινέ προκλήσεις και για τις δύο υπηρεσίες που βασίζονται και στο Γαλιλαίος και στο Κοπέρνικος. Πρώτον, έχουμε την εξάρτηση από τεχνολογία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Γαλιλαίος, αυτό αφορά κυρίως το γεγονός ότι οι περισσότερες εφαρμογές που ανατίσσονται τώρα στην αγορά βασίζονται στο σύστημα GPS. Και το δεύτερο, υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης από από εξοπλισμό που δεν έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί στην Ευρώπη. Για το κοπέρνικο, η κατάσταση είναι μάλλον διαφορετική. Ο βασικός κίνδυνος που προκύπτει είναι ότι βλέπουμε το Κοπέρνικος ως ε, άλλον πάροχο διαστημικών δεδομένων για μια ευρωπαϊκή, ε, αμερικανική επιχείρηση ε, πληροφορικής. Γιατί για να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να διχειριστούμε, να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα δεδομένα, τα τεράστιο όγκο δεδομένων που έχει ο Κοπέρνικος, ε, χρειαζόμαστε τεράστια υπολογιστική ισχύ και ισχύ αποθήκευσης. Και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι οι αμερικανικές εταιρείε πληροφορική, όπως η Google, η Microsoft και η Apple είναι πολύ πιο προηγμένες από ότι οι ε, Ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους. Δεύτερο ζήτημα, κατακαιρματισμός. Και πάλι, αν συγκρίνουμε την ευρωπαϊκή αγορά με την αμερικανική, βλέπουμε ότι εξαιτία των ζητημάτων εθνικής ασφαλείας και των εθνικών βιομηχανικών πολιτικών, η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ πιο κατακαιρματισμένη. Αν δούμε για παράδειγμα ε, τις δημόσιες προμήθειες, βλέπουμε ότι εν γέννη ε, ευνοείται ο εθνικός ανταγωνιστής. Τώρα το τρίτο στοιχείο που ανέκυψε είναι η μη συστηματική εμπλοκή των εκπροσώπων ε, του βιομηχανικού κλάδου και να προσθέσω και του τελικού χρήστη. Αυτό ίσχυε κυρίως στην αρχή, στα πρώτα βήματα ανάπτυξης αυτών των δύο προγραμμάτων, ιδίω στι στις του Κοπέρνικου. Και παρατηρούμε γενικά ότι η προσέγγιση του, της Ευρωπαϊκής Συστημικής Αρχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη κατά την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων διέπεται κατά κύριο λόγο από θεσμικές ανάγκες και όχι ανάγκες της αγοράς. Και πάλι βλέπουμε ότι ε, έτσι υπάρχει αδυναμία έναντι της αμερικανικής αγοράς, όπου συνεχώς υπάρχει το feedback ε, της αγοράς κατά την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Μετά, έχουμε προκλήσεις ε, που είναι ε, ιδιαίτερες και συγκεκριμένε για κάθε πρόγραμμα. Στο Γαλιλαίος υπάρχουν πιθανές ε, καθυστερήσεις στην εκτέλεση νέων ε, δορυφόρων. Είναι αυτό το πιο κρίσιμο. Γιατί η βάση ε, του αντίστοιχου φορέα, του αρμόδιου φορέα, το 40% του εξοπλισμού που έχει πολιθεί είναι ήδη έτοιμα για το Γαλιλαίο. Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία έχει ήδη επενδύσει σε αυτό το τομέα είναι σημαντικό λοιπόν ε, να μην υπάρξουν περαιτέρω ε, καθυστερήσεις, ε, αλλά ούτε και να αυξήσουμε τις προσδοκίες, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καλύψουμε. Από την άλλη και οι εκπρόσωποι του κλάδου από πλευρά πλοήγηση, δορυφορική πλοήγηση, αναφέρουν ότι δεν λαμβάνουν αρκετή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Κοπέρνικο έχουμε διαφορετικά ζητήματα. Τα πιο σημαντικά ήταν η πολιτική δεδομένων και πρόσβαση. Η πολιτική δεδομένα αναγκρίθηκε το 2013 και προσδιορίζει ότι υπάρχει ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, το οποίο είναι σίγουρα μια ευχάριστη εξέλιξη. Όμως η πρόσβαση δεν είναι εύκολη σε σχέση με την πρόσβαση στα δεδομένα που προκύπτουν από την αμερικανική πλευρά. Γιατί μας είπαν ότι η διεπαφή δεν είναι φιλική προς το χρήστη, τα δεδομένα είναι, ε, δεν έχουν τύχη επεξεργασίας και δεν αποθηκεύονται με αποτελεσματικό τρόπο. Άλλο πρόβλημα του Κοπέρνικου είναι το περίπλοκο σύστημα διακυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν ε, πολλοί ευρωπαϊκοί φορεί που ε, ευθύνονται για την παροχή των βασικών υπηρεσιών του Κοπέρνικου. Μέχρι τώρα, ποια ήταν η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς αυτούς τους περιορισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικά μέσα. Πρώτον, έχει στηρίξει ε, την ε, έρευνα στα διαστημικά ζητήματα. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας κατά κύριο λόγο. Θεωρούμε ότι το, το πρόγραμμα μέχρι τώρα έχει δώσει ιδιαίτερα χρήσιμα αποτελέσματα, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών του Κοπέρνικος. Ταυτόχρονα όμως μας έχουν αναφέρει οι ενδιαφερόμενοι ότι κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω για να προσαρμοστούμε περισσότερο στις ανάγκες αγοράς. Δεύτερον, νομοθετική δράση μπορούμε να εξετάσουμε ε, κανονιστικό πλαίσιο που συνδέεται με το διάστημα άμεσα και, το, και όχι. Ο ειδικό για το διάστημα ε, κανονισμός ε, θεσπίζει ένα ευρύτερο πλαίσιο, όμως τα υπόλοιπα νομοθετικά πλαίσια έχουν και αυτά ένα σχετικό παράγοντα μόχλευσης, γιατί προάγουν τεχνολογίες που ισχύουν εγκαρσίως σε όλους ή σε πολλούς τομείς που μας ενδιαφέρουν εδώ. Τρίτη κατηγορία δράσης είναι η ευαισθητοποίηση προ ε, τι επιχειρήσει, τους πολίτες και τι δημόσιες διοικησει. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε εντοπίσει τρεις πιθανές ε, κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο πολιτική. πρώτον, προτείνουμε τη βελτίωση του συντονιστικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο συγκεκριμένα, για να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό στη διακυβέρνηση των διαστημικών ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η διαστημική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στη συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Συστημική Αρχή και των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερη καθοδήγηση και αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια ενιαία προσέγγιση για μια ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανική πολιτική. Για να αντιμετωπίσουμε τους ε, περιορισμούς θα πρέπει να βελτιώσουμε τα συστήματα πρόσβασης και διανομής δεδομένων για το Κοπέρνικος, να γίνει πιο αποτελεσματικό. Δεύτερον, είναι σημαντικό να συνδυάσουμε την έρευνα, τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για να ε, ενισχύσουμε και την εμπορματοποίηση αυτών των προγραμμάτων και υπηρεσιών. Και τρίτον, περιορισμοί από πλευρά ζήτηση και πώ αντιμετωπίζονται. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε τη δημόσια διοίκηση. Υπάρχει αυτό το κλίμα αντίσταση στην αλλαγή. Και ε, μια άλλη δυνατότητα είναι να προωθήσουμε την χρήση των διαστημικών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το να κάνουμε ρητές αναφορές ε, στις δορυφορικές πληροφορίες, ε, σε μια κλαδική πολιτική, σε μια αντιστοιχή οδηγία ή με αξιοποίηση των διαστημικών δεδομένων για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα μείνω εδώ, σας ευχαριστώ την προσοχή σας και με τα χαρά να ακούσω σχόλια και ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θαυμάσια εξαιρετικά ενημερωτική συνάντηση. Τώρα θα είμαστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά στην καθημερινή δουλειά μας αλλά θα ήθελα τώρα να σημίσω από τον κύριο Τροσανόφσκι να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαστε και πλέον τόσο πολύ αριθμοί στην αίθουσα, οπότε θα συντομεύσω λίγο. τα Γκαλιλαίο και Κοπέρνικους είναι μέσα υποδομές πάρα πολύ χρήσιμες και σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή που είναι πολύτιμη. Τώρα, με δεδομένη την προσέγγισή σας και με δεδομένη με δεδομένο τον κατακαιρματισμό που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Δεν θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε τον υφιστάμενο οργανισμό GSA που έχει θέσει κανόνες ασφαλείας μεταξύ άλλων να τον χρησιμοποιήσουμε λοιπόν προκειμένου να διαχειριστούμε και τον Κοπέρνικο για τον οποίο οι παράμετροι ασφαλείας θα ήταν πάρα πολύ σημαντικές μεταξύ άλλων. Επίσης, ε, ξέρω ότι εστιαζόμαστε πολύ ε, στα θέματα της Ευρώπης, αλλά σε σχέση με το γερμανικό GPS ή το ρωσικό γκόνας κτλ. Ε, δεν θα ήταν ίσως λίγο πιο χρήσιμο να επεκτείνουμε λίγο το πεδίο για να έχουμε πρόσβαση στις αγορές των Αφρικανικών χωρών, για να δώσω ένα παράδειγμα, οι ε, η οποία πρόσβαση θα ήταν ιδιαίτερα υποφελής για τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο. Λοιπόν, πώς προωθούμε τον δημόσιο τομέα, έχουμε εκεί μια-δύο απαντήσεις αλλά πώς ενισχύουμε τον ιδιωτικό τομέα, συνοψίζοντας λέω και εγώ, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Οπωσδήποτε έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά πρέπει, θα, θα χρειαστούμε και λίγο περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε διάφορα από τα στοιχεία αυτά. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα για τις υπηρεσίες Γαλιλαίου. Η ζήτηση διέπεται ήδη από τον ιδιωτικό τομέα. Για τις υπηρεσίες παρατήρησης, γεωγραφικής παρατήρησης, δεν υπάρχει ιδιαίτερη προθυμία πληρωμής για κάποιες υπηρεσίες, όπως ένα app στο κινητό σας που σας λέει ποια είναι τα επίπεδα ακτινοβολία στην περιοχή που βρίσκεστε για παράδειγμα. Όπως το αντίστοιχο, η αντίστοιχη εφαρμογή για τι υπηρεσίε του μετρό, για παράδειγμα. Αυτό που είδαμε είναι ότι μέχρι στιγμής πρόκειται για μια ιδιαίτερη αγορά και ευθύ εξ αρχή η εμφάνιση υπηρεσιών όπως το Google Earth δημιούργησαν αν θέλετε, οριοθέτησαν τους κανόνες της αγοράς αυτής. Και η Google παρέχει πληροφορίες δωρεάν υπό μία έννοια και οι, οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να τις έχουν αυτές τις πληροφορίες δωρεάν και για αυτό είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί μια εμπορική αγορά με τέτοιου υπηρεσίε. υπηρεσίες. Για, άλλες, ε, για την πρόσβαση σε άλλες αγορές όπως η Αφρικανική όπως αναφέρατε, αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε διαρευνήσει αλλά γνωρίζουμε από την προηγούμενη, από την τελευταία έκθεση από την Ένωση Remote Sensing ιδιαίτερα για τις ε, ε πωλήσει, τις εμπορικές ε, και τις πωλήσει υπηρεσιών ε, βασίζονται σε αυτό πολλές επιχειρήσεις Τώρα αναφερθήκατε και σε έναν κατακαιρματισμό, εννοούσατε το σύστημα διακυβέρνηση ή την ίδια την αγορά. Μάλιστα, το σύστημα διακυβέρνηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί πολύ και έχει, δημιουργεί, έχει οδηγήσει σε μεγάλες διαφωνίε. Στην περίπτωση του Γκαλιλαίου έχουμε έναν οργανισμό αυτόν τον, δορυ... τον οργανισμό δορυφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τη χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τον Κοπέρνικο αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να είναι μια επιλογή που θα, εξε... θα έπρεπε την ανάπτυξή της. Σας ευχαριστώ αγαπητοί Τελπόντε για την παρουσίασή σας καθώς και τις χρήσιμες συμβουλές σας για το πώς να κινηθούμε και από την ε, άποψη βέβαια δική μας ως πολιτική, διότι <clears throat> είπατε τρία πράγματα στο τέλος. Ένα απλό για μας τους πολιτικούς και ασφαλώς το λαμβάνουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία μου. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Debriefing και feedback από τους συντονιστές. Τουλάχιστον να με ακούσετε εσείς βοηθή αφού όλοι οι ευρωβουλευτές απεχώρησαν. Πάντως εξακολουθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ενέργειας. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι παρόν. Λοιπόν, New Energy Market Design, 17 Μαρτίου. Ακρόαση, πολύ σημαντική ακρόαση. 17 Μαρτίου, ξαναλέω. New Energy Market Design. Ακρόαση, ξαναλέω, πολύ σημαντική. καταχώρησης, το GPS, αυτό το τελευταίο που ακούσαμε κιόλας, μεταξύ χωρών μελών και νιανιά, ε, η ομάδα ENF. Τέσσερα, τέσσερις, τέσσερα άλλα σημαντικά νομοθετήματα, κυκλική οικονομία. Οικονομία και τέλος ζωής διάφορων αναλώσιμων μπαταρίες κλπ. Στην άλδε κυκλική οικονομία, πάλι ε, ε, χώροι ε, ταφής απορριμμάτων. Άλντε. Πάλι S&D για το τρίτο αυτό του πακέτου και τέταρτο που είναι οι ε, ε συσκευασίες ε, στην ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Τώρα τα γνωρίζετε όλα. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2016 βέβαια, το απόγευμα της 22ης και το πρωινό και απόγευμα της 23ης Δευτέρου 2016. Σας ευχαριστώ πολύ και σας απολύω.